Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τη συνεδρία της Επιτροπής μας και περνάμε στο σημείο 11 της ημερήσια διάταξης. Στο εξή 10. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ο Καλχάινς Φλόρενς είναι ο εισηγητής μα, εξαιρετικό, όχι είναι το 11 θέμα τελικά, και θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Φλόρεντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 2002 Το 2002 για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή προσπαθήσαμε να περιορίσουμε και να οργανώσουμε ε, τα, ε, της διαχείρισης των αποβλήτων ε, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού ε, εξοπλισμού. Ήταν μεγάλη υπόθεση ε, μετά τα αυτοκίνητα. Προσπαθήσαμε να συμπλησιάσουμε τους κανόνες και το δίκαιο, γιατί ξέρουμε ότι το δίκαιο για τα απόβλητα μπορεί να καθορίζεται στο πλαίσιο του από τις Βρυξέλλες, αλλά η εφαρμογή σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τα κράτη-μέλη, γιατί εκεί υπάγεται και από την πρώτη οδηγία είχαμε πολύ περίεργα πράγματα που προέκυψαν τελικά, διότι ήταν τελείως νέο το πεδίο και ο κόσμος δεν ήξερε πάρα πολύ καλά πώς μπορούν να εφαρμοστούν όλα στην πράξη. Επίσης υπάρχουν και καινούργια θέματα που έπαιξαν ρόλο πριν από λίγα χρόνια και τελικά δεν ξέραμε πώς θα τα εφαρμόσουμε όλα αυτά. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα ηλεκτρονικά απόβλητα έχουν γνωρίσει τεράστια αύξηση σε όγκο τα τελευταία χρόνια και στο μέλλον θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Αν δεν το πιστέψετε, κοιτάξτε στο σπίτι σας τι γίνεται και αν έχετε και παιδιά, τι συσκευές και πόσες έχετε αγοράσει και πόσο γρήγορα παλιώνουν. Γι' αυτό ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ ε, αυτές οι πρώτες ύλες ε, να ε, αποσύρονται σωστά, να ε, βγαίνουν τα δηλητήρια που έχουν μέσα και να ανακυκλώνονται. Και η ιδέα ήταν λοιπόν γύρω στο 2000 πολύ ρηξικέλευτη, γιατί ήδη από τότε ξέραμε ή υποπτευόμαστε ότι στο μέλλον θα σπάνιζαν ακόμα περισσότερο οι πρώτες ύλες και αυτή η οδηγία μας βοηθάει καλύτερα να αντιμετωπίσουμε τη σπάνη των πρώτων υλών. Και έρχομαι τώρα στο μελλον θα σπανιζαν ακομα περισσοτερο οι πρωτες υλε και αυτη η οδηγια μας βοηθαει πρόβλημα που δυστυχώς ε, ερχόμαστε να διαπιστώσουμε ότι στην πρώτη οδηγία δεν είχαμε πετύχει πάρα πολύ, δεν τα καταφέραμε τόσο καλά όσο θα επιθυμούσαμε, διότι μόλις 40% των ηλεκτρονικών συσκευών στο λιανικό εμπόριο ε, μπήκαν σε αυτή την οδηγία μόνο το 40% και τελικά ερχόμαστε να διαπιστώσουμε ότι δεν είναι παραπάνω από 33% όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που πέρασαν από αυτό το κανάλι. Τώρα θέλετε μπορούμε να διαπληκτιστούμε γιατί είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό. Τελικά όμως και αυτό είναι κρίμα, 70% δεν ρυθμίζεται. Ε, δηλαδή δεν είναι σαφές τι γίνεται με τα ε, ε, υγρά, τα αέρια, τα επικίνδυνα, τα τοξικά που μπορεί να βλάπτουν και την υγεία. Πού πηγαίνουν όλα αυτά που είναι μέσα στις συσκευέ. Δεν τα πετάμε όλα έτσι όπως να είναι στη χωματερή, προφανώς. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη φαιά ζώνη εκεί και σκοτεινά σημεία και καλό είναι να ασχοληθούμε με αυτό. Και επίσης είναι σωστό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέδρασε και μας έκανε κάποιες προτάσεις πολύ ενδιαφέρουσες και ελκυστικές. Βέβαια πάντα υπάρχουν κάποιοι που είναι αντίθετοι με αυτές τις ρυθμίσεις. Έχουμε τεράστια ενιαία αγορά και γι' αυτό ήρθα εγώ στην Ευρωβολή και όχι στη Βουλή της χώρας μου, στην Bundestag και ακριβώς ε, σε αυτό το κλάδο δεν θα πρέπει να ε, το βλέπει ο καθένα στη χώρα του εθνικά να το ρυθμίζει. Ε, νομίζω ότι πρέπει να το ξανασυζητήσουμε αυτό. Έρχομαι λοιπόν τώρα στι λεπτομέρειε. Πρώτον, και ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην παλιά οδηγία και στι παλιέ ρυθμίσει και στον παλιό κανονισμό λέει ότι το πεδίο εφαρμογή ε, στα δύο έγγραφα, το Β και το Ρος, τα ξέρουν οι συνάδελφοι, θα Ε, ρυθμιστούν στο, στο V έλεγε το πρώτο, το electronic waste δηλαδή. Και τώρα όμως θα μπουν στο ροζ, αν κατάλαβα καλά. Ε, ε, στο label 95. Δεν ξέρω ποιες είναι οι διαγραφές και τι λέει η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Το θέμα είναι όμως πού θα βάλεις τις προδιαγραφές. Αν είναι ψηλά ο πύχης, εντάξει, συμφωνώ με το 95. Αν είναι όμως χαμηλές, οι απαιτήσει όχι. Παρακαλώ να το κοιτάξει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί το πρώτο είναι έτσι, γιατί θα πρέπει η ρύθμιση τώρα να έχει το πεδίο εφαρμογή στο ΡΟΥΣ. Γιατί δεν παραμένουν τα δύο θέματα ξεχωριστά Γιατί η ποσόστοση ε, Άλλοι λένε 5 κιλά, άλλοι λένε 11 κιλά, ε, άλλοι λένε καθόλου να μην βάλουμε, οι πιο πονηροί, στο ΙΤΕΣ. Τα είπε πολύ ωραία η κυρία Μακάβαν το πρωί. Το ίδιο ισχύει και ε, ε, με το φάκελο αυτό. Έγινε μεγάλη φασαρία στα τρία θεσμικά όργανα και καταλήξαμε στα τέσσερα κιλά. Γιατί ήταν δύσκολο για τις νέες χώρες να βάλουν πιο ψηλούς ε, αριθμούς και να τους στηρίσουν. Τότε, ε, ήδη από τότε η Γερμανία είχε 14-15 κιλά και η Αυστρία. Τελικά καταλήξαμε στα 4 σε συμβιβασμό. Τώρα θέλουμε να το αλλάξουμε. Δεν θα βάζουμε κιλά, θα βάζουμε ποσοστά. Και τα ποσοστά αυτά θα πρέπει να προσανατολίζονται ε, στα δύο τελευταία έτη πωλήσεων ε, από την κυκλοφορία ενός προϊόντος στην αγορά. Βέβαια μπορούμε να τα συζητήσουμε αν θέλετε και τα ποσοστά, αλλά παρακαλώ δεν ε, θεωρείται αυτό ποινή ή τιμωρία το ποσοστό. Με τα ποσοστά θέλουμε να εξασφαλίσουμε τις πρώτες ύλες για τα εγγόνια και τα δυσέγγονά μας. Δεν θέλουμε να αγοράζουμε προϊόντα, να τα χρησιμοποιούμε, να τα πετάμε ή λαθρέα να τα εξάγουμε κάπου και να τα πετάμε αλλού, αλλά θέλουμε εξοικονόμηση πρώτων υλών και ανακύκλωση. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι οι στόχοι μας στα ποσοστά φιλόδοξη. Στα νέα κράτη-μέλη μπορεί να υπάρχουν έτσι εδώ αντιστάσεις και προβλήματα, το κατανοώ αυτό και το δέχομαι. Αλλά κάποια λύση θα βρούμε. Εδώ λοιπόν ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει σήμερα υψηλή εκπροσώπηση, πώς καταλήγετε σε αυτό το 65% παρακαλώ, μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Και ελπίζω να ε, κάνετε προτάσεις ε, business to business και business to customer, to consumer. Μπερδεύεται λίγο μιλητής και κάνει και σαρδά. Λοιπόν, είναι πολύ φιλόδοξη η πρόταση. Ε, χαμός έχει γίνει στο γραφείο μου από πιέσει. Και θέλω να ρωτήσω επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα γίνει μέχρι το 2016, γιατί αυτά που προτείνει, λέει, θα τεθούν σε ισχύ το 2016. Ε, στο μεταξύ όμως τι θα κάνουμε. Δεν υπάρχει κενό εδώ. Και πώς θα καλυφθεί ενδεχομένω. Ε, δεν ξέρω, σταδιακή ρύθμιση, βαθμιαία. Είπα προηγουμένως ότι μόνο 30% περνάει από το triple E ε, κανάλι στην ανακύκλωση ή στην διάθεση, την τελική, αλλά θα πρέπει να ορίσουμε πάρα πολύ ξεκάθαρα πού θα πρέπει να υπάρχουν αυτά, αυτές οι συσκευές, ποιος να πληρώνει μέχρι πότε. Ορισμένοι λένε ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Άλλοι λένε ότι ακόμα και μια ηλεκτρική οδοντόβορτσα να έχει θα πρέπει να πάνε να την πάρουν από το μπάνιο. να έρθουν να την πάρουν από το σπίτι του και όχι να πάει εκείνος να την πετάξει κάπου. Και ο χρήστη θα πρέπει να έχει μια κοινωνική ευθύνη και ένα αίσθημα καθήκοντος σε πάση περιπτώσει, να πηγαίνει και αυτός ε, τη συσκευή σε κάποια θέση συγκέντρωση αυτών των αποβλήτων ή ε, να το ρυθμίζουν οι χώρες ε, πώς θα γίνεται η παραλαβή αυτών των συσκευών. Για να μην χάνονται στο δρόμο. Δεν ξέρω τι γίνεται στις χώρες σας κυρίες και κύριοι. Άμα βγάλει κανείς στη Γερμανία ένα ψυγείο 8 η ώρα το βράδυ, την άλλη μέρα το πρωί 8 έχει εξαφανιστεί το ψυγείο. Όχι ότι το μαζεύουν τίποτα επίσημοι, αλλά ρακοσυλέκτες δεν έχω πρόβλημα, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται με αυτό το ψυγείο. Τι θα γίνει με τα υγρά, τα επικίνδυνα που έχει μέσα το ψυγείο. Ποιος θα τα ε, βγάλει αυτά και θα το καθαρίσει. Έτσι. Δεν είναι καθόλου εύκολα αυτά, το καταλαβαίνω, αλλά το 33% θα πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθεί. Δεν μπορεί να χάνονται οι υπόλοιπε συσκευέ από αυτό το κύκλωμα θα πρέπει να μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έρχομαι τώρα ε, στην πιο δύσκολη για μένα ερώτηση, που είναι η καταχώρηση των ε, κατασκευαστών και ορισμός αυτής. Και πάλι είχε γίνει μεγάλη φασαρία και καυγά τότε, γιατί θέλαν όλοι οπωσδήποτε να τα ρυθμίζουν εθνικά τα πάντα, σε επίπεδο κράτους μέλους. Και στη δική μου χώρα, ε, εκεί που ζω, θέλω να το κάνουν στα 16 ομόσπονδα κράτη και στην Αυστρία τα ίδια. Οι Γερμανοί τουλάχιστον κατάφεραν να το ρυθμίσουν εθνικά σε ένα επίπεδο και όχι σε 16. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η καταπληκτική και σπουδαία εσωτερική αγορά κανονικά θα πρέπει να είναι σε θέση να έχει ένα μητρό, μία δυνατότητα καταχώρησης για όλους. Α είναι ο καθένα στη χώρα του, δεν με νοιάζει αυτό, ε, όπου εδρεύει κάθε χώρα, αλλά κάπου, η κάθε εταιρεία, συγγνώμη. Αλλά κάπω μετά να υπάρχει μια διασύνδεση, μια ενημέρωση έτσι ώστε να ξέρουμε ότι ένα πλυντήριο που επιτρέπεται να κυκλοφορεί στην Ολλανδία να αγοράζεται και στην Πορτογαλία, για παράδειγμα. Μεγάλες αντιστάσεις εδώ, τρομερές. Και μας κάνει εντύπωση ότι φωνάζουν αυτοί που φωνάζουν συνήθως για τη χρηματοδότηση. Αλλά, πώς να το πω, δεν θα πρέπει να αφήσουμε να μας παραπλανήσουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Έχουμε ενιαία αγορά, μία. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι η διαχείριση ανάμεσα στο Βερολίνο και στο Μόναχο είναι πιο δύσκολη από ότι ανάμεσα στο Βερολίνο και την Πορτογαλία. Καμιά φορά είναι πιο απλό να συνεννοηθεί το Βερολίνο με την Πορτογαλία παρά με τη Βαβαρία. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποια είναι η δυνατότητα ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εάν από εκεί και πέρα στην καταχώρηση στις άδειε αναπτυχθεί η αγορά, έτσι, δεν είναι και κακό να είναι κάπου πιο ψηλές οι προδιαγραφές, είναι κίνητρο. Για μένα θα ήταν τρομερή οπισθοδρόμηση εάν οι αρμόδιες αρχές, και εδώ ανήκει και το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Γερμανίας, αλλά και πολλοί άλλοι θεσμοί που ασχολούνται με την πραξή των εσόδων ενός κράτους, θέλουν να διατηρήσουν τα κεκτημένα και το καθεστώς, το καταλαβαίνω. Αλλά να κάνεις 27 διαφορετικούς οργανισμούς για αυτό το πράγμα, μου φαίνεται πολύ μεγάλη πολυτέλεια. Και για την εθνική οικονομία, τα πανηρότατο. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί άλλη λύση. Ένα μόνο οργανισμό χρηματοδότησης πάλι δύσκολα το βλέπω να γίνεται. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις της βιομηχανίας. Για μένα είναι πολύ παλιωμοδίτικες και δεν μπορώ καν να τις υποστηρίξω. Μέχρι τώρα υπήρχε ένας χώρος συγκέντρωσης και αυτό ήταν το αποφασιστικό για το πού θα αναλάβει το κόστος ο παραγωγός, ο κατασκευαστής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να είναι στην πόρτα του νοικοκυριού. Εντάξει, ας το δεχτώ και αυτό. Παρόλο που προσωπικά έχω άλλη άποψη. Θα πρέπει και ο καταναλωτή λίγο να έχει μια ευθύνη και μια ευαισθησία να πηγαίνει ο ίδιο στη συσκευή του κάπου. Εν πάση ε, αυτά ήθελα να σας προτείνω. Αυτά είναι τα σημαντικότερα. Έχουμε μια ειδική διαδικασία που δεν μπορώ να την προφέρω, δεν είναι επιτροπολογία, μια άλλη πώς τη λένε. Κάποτε αποφασίσαμε, κύριε Πρόεδρε, ότι εμείς έχουμε δικαίωμα να αντιδράσουμε μόνο σε ό,τι θεωρεί σωστό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας προτείνει να αλλάξουμε. Αν είναι δυνατόν. Εγώ πάντα θεωρούσα ότι το Κοινοβούλιο ελέγχει τη δίκηση. Μου φαίνεται έχω μείνει πίσω και <laughs> πρέπει να αλλάξω μυαλά. Όταν ένα κοινοβούλιο θεωρεί ότι κάπου πρέπει να παρεμβαίνει κοινοβουλευτικά, πρέπει να το κάνει. Τι είναι αυτή η διαδικασία που επιλέξαμε, ότι μπορούμε δηλαδή να αντιδράσουμε μόνο στους τομείς που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητήσουμε, γιατί θεωρεί εκείνη ότι χρειάζεται αλλαγή. Για φαντάσου. Εκείνη τη μέρα εγώ το υπερψήφισα αυτό. Ε, δεν ήμουν και στο φόρτε μου φαίνεται. Θα ήθελα να μας πει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τον ορισμό τι είναι το business του, business και business του consumer και το θέμα της έγκρισης και τα οικονομικά συστήματα, όλα αυτά νομίζω ότι είναι φρικτή γραφειοκρατία στην Ευρώπη χωρίς ε, καμία έννοια της αγοράς και της ε, οικονομίας της αγοράς. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε εκεί χρήματα και να τα βάλουμε στο περιβάλλον πολύ πιο χρήσιμα αλλού. Ευχαριστώ πολύ, Καρλ Χάινς Φλόρενς, για την ε, πολύ καλή αυτή εισαγωγή στο θέμα. Στην ε, επόμενη σύνοδο θα μπορέσετε να απαιτήσετε να γίνουν τα πράγματα όπως θέλετε. Το Κοινοβούλιο πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει ε, το δικαίωμα της πρωτοβουλίας ούτε με την ε, νέα συνθήκη. Ζητήσατε από την Κομισιό να απαντήσει σε κάποια θέματα. Παρακαλώ τον Κλάους Κίκλερ από την Κομισιό να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για τις αρχικές αυτές παρατηρήσεις. Καλό απόγευμα σε όλους. Να ξεκινήσω από το τελευταίο θέμα που ανέφερε ο κύριος Φλόρενς, γιατί επιλέξαμε τη ε, διαδικασία της αναδιατύπωσης. Αυτό δεν έγινε για να μην συμμετάσχουν άλλα θεσμικά όργανα στη συζήτηση. Το κάναμε καλή την πίστη ιδιαίτερα επειδή η διαδικασία ε, αναδιατύπωσης αποτελεί χρήσιμη μέθοδο κατά την αναθεώρηση μιας τόσο ε, ενός τέσου νέου νομοθετήματος. Κατά την αναδιατύπωση πάντα υπάρχει κάποια ανασφάλεια και ανησυχία. όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια θέση και η διαδικασία της αναδιατύπωσης προστατεύει κάποιες ρήτρε που δεν φαίνεται να χρειάζονται αναθεώρηση. Η διαδικασία της αναδιατύπωσης λοιπόν επιλέγει, έχει επιλεγεί για να διασφαλίσει κάποια συνέχεια και στη διοίκηση και για τους οικονομικούς φορείς που πρέπει να συνεχίσουν τις εργασίες τους ενώ εμείς διαπραγματευόμαστε πιθανές βελτιώσεις. Ποιο ήταν το σημείο κίνησης κατά τη συζήτηση της πρότασης αυτής. Η κατάσταση ήταν αρκετά απλή. Είχαμε ένα σχετικά νέο νομοθέτημα για το οποίο συλλέξαμε ε, κάνα δύο χρόνια μόλις πρακτικής εμπειρίας. Ο εισηγητής νομίζω ανέφερε με πολύ πλήρη τρόπο κάποια τεχνικά διοικητικά θέματα που προέκυψαν και που η πείρα έδειξε ότι χρειάζονται επανεξέταση. Από περιβαλλοντικής πλευράς διαπιστώσαμε ότι τα τοπικά μέτρα δεν ανταποκρίνονταν στη φιλοδοξία της, στις φιλόδοξες προθέσεις της οδηγίας. Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στην πρόταση αυτή να επανέλθω στις ερωτήσεις. Γιατί προτείνουμε να αλλάξουμε την σειρά στην παρούσα κατάσταση όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής η μία οδηγία προτείνει το πεδίο εφαρμογή και η άλλη το ακολουθεί. Αυτό αποτελεί λίγο ένα πρόβλημα, διότι ε, η οδηγία ΡΟΣ είναι του 95 και είναι αρκετά δεσμευτική. Εάν έχουμε μία μη δεσμευτική οδηγία, αυτό οδηγεί σε ανασφάλεια και σε μπέρδεμα. Προσπαθήσαμε λοιπόν να λύσουμε το πρόβλημα αντιστρέφοντας την κατάσταση. Στη νέα μας πρόταση λοιπόν, το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει έναν ελάχιστο δεσμευτικό κατάλογο προϊόντων που είναι εξαντλητικός για την οδηγία ΡΟΣ. Εκεί δηλαδή το πεδίο εφαρμογής είναι σαφές. Και αυτό αποτελεί το ελάχιστο πεδίο, το μπορεί όμως αυτό να τροποποιηθεί ανα πάσα στιγμή, σύμφωνα με το άρθρο 95. Επίσης, ρωτήσατε μήπως θα έπρεπε να διασφαλίσετε ένα υψηλό επίπεδο ε, προτύπων προστασίας. Δεν νομίζουμε ότι το να καθορίσουμε το πεδίο εφαρμογής ως προς τα προϊόντα που καλύπτονται ε, εμποδίζει να γίνει κάτι τέτοιο. Η δεύτερη ερώτηση είχε να κάνει με το στόχο. Ο στόχο όπως τον παρουσιάζει η Επιτροπή είναι λογικό από πού προέρχονται τα ε, στατιστικά στοιχεία. Εν μέρη από ό,τι γνωρίζουμε ήδη έχετε αναφέρει τα στοιχεία αυτά. Το 85% των ε, προϊόντων ε, που προκύπτουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση συλλέγεται σήμερα και αυτό ουσιαστικά μεταφράζεται στο 65% των όσων έχουν διατεθεί στην αγορά τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς, από το 85% αυτό ε, δεν έχουμε πολλά στοιχεία από τα κράτη-μέλη και αυτό οδηγεί σε μια σημαντική ανησυχία ότι μέχρι και το 55% πιθανότατα μπορεί να ε, αποτελεί αντικείμενο παράνομης ε, διαχείρισης, ε, διαχείρισης που να μην πληρεί τα κριτήρια και στη χειρότερη περίπτωση παράνομες εξαγωγές. Ακούσαμε την αιτιολόγηση, τη διασφάλιση δηλαδή των πρώτων υλών, αλλά και τη διασφάλιση της σωστής διαχείρισης, της σωστής διάθεσης Ε, φροντίζουμε το 85% που συλλέγεται να ε, διατίθεται σύμφωνα με τα πρότυπα. Το 85% δηλαδή που, που προκύπτει που αντιστοιχεί στο 65% των προϊόντων που διατίθεται στην αγορά. Πιστεύουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε κάτι τέτοιο. ρωτήσατε ως προς την ε, συλλογή ε, αν θα πρέπει να ε, διευρύνουμε την υποχρέωση του πολιτή να συλλέγει τα προϊόντα από την πόρτα του καταναλωτή. Πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί υπό όρους να βοηθήσει τους καταναλωτές να πληρούν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την συλλογή των, του παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Διότι κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει ένα αίσθημα ιδιοκτησία στους παραγωγούς εάν ε, είναι υποχρεωτικό. Ωστόσο, δεν το κάναμε αυτό υποχρεωτικό, διατηρήσαμε τη διάταξη όπως είναι ήδη διατυπωμένη σήμερα, ότι αυτό μπορεί να γίνεται, δεν είναι όμως υποχρεωτικό. Ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να εξετάσουν αυτή την, την εναλλακτική αυτή λύση, ε, αλλά δεν είναι υποχρεωτική από την πλευρά μας ως προς τους καταλόγους στα Μητρώα. Αυτό ήταν το δεύτερο σημαντικό θέμα κατά την αναθεώρηση και ο τομέας που χρειαζόταν ε, βελτίωση. Πριν δύο-τρία χρόνια, κατά τη διάρκεια διαβουλεύσεων, όταν ακούσαμε τους οικονομικούς φορείς και άλλους ενδιαφερομένους, ε, ένα πρόβλημα που ανέκυπτε ήταν το απαράδεκτο ε, επίπεδο διοικητικού φόρτου λόγω του ότι οι οικονομικοί φορείς έπρεπε να κάνουν πολλαπλή καταχώρηση σε, σε πολλές χώρες. Συχνά έπρεπε μάλιστα να καταβάλουν πολλαπλά τέλη για τον ίδιο εξοπλισμό. Θέλαμε λοιπόν ένα μητρό το οποίο να πληρεί κάποια ελάχιστα κριτήρια απλοποιημένης λειτουργίας. Ε, η πρώτη αυτή απέτηση ήταν μία καταχώρηση, μία αίτηση ή μία ηλεκτρονική αίτηση σε κάθε ένα από τα 27 κράτη-μέλη θα πρέπει να αρκεί και οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να διαβιβάζονται σε όλα τα άλλα Και έτσι ο οικονομικός φορέας να ε, έχει τελειώσει τη δουλειά που πρέπει να κάνει από τη μεριά του. Αυτή λοιπόν η μία και μοναδική καταχώρηση θα πρέπει να επιτρέπει την ε, καταχώρηση σχετικά με τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρονικά προϊόντα που διατίθεται στην αγορά σε κάθε ένα από τα κράτη-μέλη. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται και ενημέρωση άλλων μητρών σχετικά με πιθανές ε, διπλές πληρωμές. Θα οδηγήσει δηλαδή σε αποφυγή διπλών τελών θα πρέπει να είναι δυνατή κάποια πληροφόρηση σχετικά με τη ροή χρημάτων, δηλαδή μέσω του συστήματος αυτού. Επίσης θα θέλαμε να βρεθούμε στην κατάσταση όπου δεν θα είναι απαραίτητο για έναν οικονομικό φορέα να έχει νομική έδρα σε κάθε κράτος μέλος το οποίο δραστηριοποιείται. Πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες λύσεις που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε. Με τις πρώτες αυτές παρατηρήσεις ελπίζω να απήντησα στα βασικά ζητήματα σας κύριε εισηγητά και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις σε περίπτωση που ξέχασα κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κίκνερ για τις πληροφορίες αυτές. Μέχρι τις 4 έχουμε χρόνο και έχω 8 ομιλητές. Εάν δεν θέλει να μιλήσει κανένας άλλος, να κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Ωραία. Τρία λεπτά το πολύ τότε. Δέκα ομιλητές έχουμε τώρα. Δύο με τρία λεπτά. Παρακαλώ. Κυρία Βαν Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομη εγώ. Δεν είμαι νέα στο Κοινοβούλιο. Πριν από έξι χρόνια πέρασα κι εγώ ένα διάστημα και τότε είχα ασχοληθεί με πάθος με αυτό το θέμα. Έτσι δεν είναι, Καλχάιντ, θυμάσαι. Και χαίρομαι που και πάλι το ε, ανέλαβα. Είναι πολύ σημαντική η οδηγία. Άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέγει ότι αξίζει να αναθεωρηθεί και να βελτιωθεί σίγουρα η οδηγία. Αν μπορούμε να προχωρήσουμε σε διοικητικέ απλουστεύσεις για τα κράτη-μέλη, τόσο το καλύτερο. Και ε, αν ε, θέλουμε να πετύχουμε και τους περιβαλλοντικούς στόχους, επίσης είναι καλό. Βέβαια, να δούμε με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα χρειαστούν ε, συζητήσεις γι' αυτό. Για το πεδίο εφαρμογής νομίζω είναι καλή η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρειάζεται λίγο περισσότερο ψάξιμο. Επειδή δεν έχω και πολύ χρόνο, θέλω να τονίσω τα εξή. Εξεπλάγει πάρα πολύ από αυτό που μας είπε τώρα μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το στόχο του 65%. Η αρχική μου ιδέα ήταν ότι το 65% είναι καλό να παραμένει σχετικό στόχος και όχι απόλυτος, κατά κεφαλή. Εντάξει, καλό βήμα αυτό, αλλά το βρίσκω και πολύ περιορισμένο. Και η απάντηση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εκπλήσει. 85% των συσκευών, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση συλλέγονται σωστά, αλλά μετά δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Δηλαδή, αυτό το 65% πες ότι μπήκε ο στόχος. Είναι φιλόδοξος. Αλλά ίσως θα πρέπει να βάλουμε περισσότερους στόχους ε, για πιο απότερο διάστημα. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο να μαζεύουμε τις συσκευέ, αλλά να έχουμε καλύτερο έλεγχο και επιθεώρηση από εκεί και πέρα τι γίνεται. Για να φροντίσουμε όλοι μας να ενισχυθεί η οδηγία και να εφαρμόζεται σωστά. Δεύτερο, είναι πιο μακροπρόθεσμα και ήταν από τα θέματα που με απογοήτευσαν στην αρχή ακόμα της πρότασης αυτή και με πίκραναν ήταν ότι υπήρχε η ευθύνη του κατασκευαστή ως αρχή. Εντάξει, το έγραφε αυτό η οδηγία, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη. Δηλαδή δεν διατυπώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε στην πράξη να επιβληθεί. Έχουν περάσει τα χρόνια βέβαια. Είναι υπεύθυνοι κατασκευαστές και βγάζουν καλά προϊόντα, εντάξει, αλλά ε, και αυτό πρέπει να βελτιωθεί. Όχι μόνο οι μεμονωμένοι λοιπόν κατασκευαστές και οι διευθύνοι του για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά να δούμε πώς ανακυκλώνονται, πώ συλλέγονται και πώ χρησιμοποιούνται τελικά. Και να είναι και πιο καλά τα προϊόντα. Ξέρετε και την περίφημη αρχή cradle to cradle, ε, ε, ένας πολύ διάσημος γερμανός ε, καθηγητής την είχε φεύρει, Δηλαδή από την γέννηση ενός προϊόντος μέχρι τη γέννηση του επομένου προϊόντος. Αυτά. Ελπίζω να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την οδηγία. Η δική μας πολιτική ομάδα σίγουρα θα σας υποστηρίξει στη στόχευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θεώρηση οδηγίας. Ευχαριστώ. Υπάρχουν συνάδελφοι που αγαπούν τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Δεν μπορούν να το αφήσουν αυτό το θέμα. Συναρπαστικό ο κλάδο. Ε, είναι δραματικέ οι αραγέ. Ο κύριο Παναγιώτοφ, παρακαλώ. Σα Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το πολύ σημαντικό θέμα θα ήθελα να το τονίσω ακόμη περισσότερο, διότι πρόκειται για νέους πόρους, νέους πόρους για την Ευρώπη. Πώς θα μπορέσουμε να βρούμε νέες δυνατότητες για να έχουμε στρατηγικά στοιχεία για την Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη πληρώνει, δίνει πολλά χρήματα κάθε χρόνο για να διατηρήσει αυτά τα, τα ηλεκτρονικά, τι ε, ηλεκτρονικές συσκευές, στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν που πρότεινε το θέμα γιατί είναι εξαιρετικά πολύτιμο. Στόχος είναι να δούμε πώς θα μπορέσουμε με τον καλύτερο τρόπο να ανακτήσουμε αυτά τα στοιχεία να δείξουμε πως είναι πολύ ωφέλιμο για μας, να το παρουσιάσουμε για τις 27 χώρες και να εφαρμόσουμε αυτού του είδους τη νέα τεχνολογία τη νέα ε, νοοτροπία, διότι αυτό είναι ευκολότερο ευκολότερος είναι ευκολότερος για μας, παρότι δεν είναι εξαιρετικά εύκολο, αλλά τα ηλεκτρονικά κατάλοιπα βοηθούν στο να ανακτηθούν πολλά πολύτιμα στοιχεία. Ευχαριστώ κύριο Στρεμόπουλος, παρακαλώ. No? Then, uh, Julie um, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Γκέρλινγκ. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες αρχικές παρατηρήσεις από πλευράς της ομάδας μου. Διαβάζοντας ε, την προτινόμενη αναθεώρηση από την Κομισιόν, με εντυπωσίασε αυτό που εγώ θεωρώ έλλειψη ε, ε, ενημέρωσης όσον αφορά την κατανόηση της αγοράς ε, καταναλωτή. Εγώ περίμενα ότι θα αυξηθούν τα επίπεδα τα οποία αφορούν την ανάκτηση υλικών. Τίποτα δεν μας λέει εδώ γιατί ορισμένοι τομείς θα πάνε καλύτερα και ποια προϊόντα ανακυκλώνονται σε ψηλότερο ποσοστό. Ε, φαίνεται να υπάρχει μεγάλη παρανόηση της αγοράς. Ε, έχουμε πολλά πολλά στοιχεία, ε, αλλά δεν ξέρουμε πού δεν ανταποκρίνεται η συμπεριφορά των καταναλωτών και των ε, πολιτών στην επιθυμία μας. Εδώ δεν θέλουμε να μιλήσουμε μόνο για τον κανονισμό, αλλά για το πώς θα κάνουμε τους παραγωγούς και τους ε, πολίτες, τους καταναλωτές, να ασχοληθούν και να συμφωνήσουν και να προσπαθήσουν και για τους δικούς μας στόχους. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο δεν έχει τίποτα που να λέει πού πάνε καλά τα πράγματα και πού μπορούμε να βελτιώσουμε. Υπάρχει ένας αυθαίρετος αριθμός 65% ε, που όμως δεν μας βοηθά να καταλάβουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πώς θα μπορέσουμε να κρίνουμε αν αυτή η αναθεώρηση έχει λειτουργήσει. Είναι η ευκαιρία μας να το φτιάξουμε έτσι ώστε να μπορούμε να παρακολουθήσουμε την αποτελεσματικότητα. Πράγμα που δεν μπορέσαμε να κάνουμε με τον αρχικό κανονισμό. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες γιατί δεν έχουμε αρκετές για να μπορέσουμε να κρίνουμε. Ευχαριστώ πολύ ο Ρίχαρτ Σίβερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν για τις παρατηρήσεις τους. Και εγώ πιστεύω σε μια ευρωπαϊκή στρατηγική πόρων που θα συμπεριλαμβάνει μια, την ανακύκλωση των, ε, του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Δεν κατάλαβα πολύ καλά αυτά που είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν σχετικά με την ε, νομική μορφή. Γιατί θα πρέπει να είναι αναδιατύπωση. Ε, εμείς θα πρέπει να αποφασίσουμε κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι η επιλεγμένη μορφή δεν είναι η σωστή και δεν είμαι ικανοποιημένος. Επίσης πιστεύω ότι η νομική βάση που έχει επιλεγεί δεν είναι η σωστή. Πιστεύω ότι το άρθρο 95 θα ήταν καλύτερη νομική βάση και όχι μόνο το άρθρο 175. Δεύτερον, βλέπω να υπάρχουν προβλήματα επειδή υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό το 65% που θέλουμε να πετύχουμε είναι δύσκολο να επιτευχθεί λόγω των μεγάλων διαφορών που υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών. Θέλουμε να εισάγουμε τον όρο του Ευρωπαίου παραγωγού με την πρόταση αυτή, αλλά πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα σχετικά με την εφαρμογή του νόμου. Δυστυχώς η εσωτερική αγορά υποφέρει από τα διαφορετικά συστήματα εφαρμογής που υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή προχωράει σωστά προς την εσωτερική αγορά, ε, δεν αρκούν όμως τα βήματά της. Το πρόβλημα λοιπόν είναι η σωστή εφαρμογή του νόμου και κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Στην παλιά οδηγία έχουμε τα εθνικά συστήματα, τα οποία πότε λειτουργούν καλά, πότε όχι. Αλλά κατά τη γνώμη μου η επιλεγμένη προσέγγιση ήταν αρκεί. Και επίσης θα πρέπει να γίνει η κατανομή των αρμοδιοτήτων και του φόρτου μεταξύ, ανάμεσα στους ε, παραγωγούς και στους καταναλωτές. Υπάρχουν τα συστήματα συλλογής και αξιολόγησης και ε, ε, ε, ανακύκλωσης. Λειτουργούν συνήθως σε δημοτική βάση στα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι στην οδηγία θα πρέπει να διευκρινίσουμε πώς θα λειτουργήσουν αυτά στο μέλλον. Τον διακόπτει ο πρόεδρος τον ομιλητή. Τρία λεπτά έχετε. Εντάξει κύριε πρόεδρε, σταματάω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζήπερ. Ο Βιτόριο Πρόντι. Grazie Presidente. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να αναφερθώ στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα που προβλέπει την ε, εκ νέου χρήση, την ανάκτηση, την ανακύκλωση και την καταστροφή με τη σειρά. Δεν βλέπω λοιπόν πώς εδώ έχουμε προσπαθήσει να πάμε μπροστά σε αυτή την οδηγία, προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, η χρήση εκ νέου τόσων μηχανών, τόσων μηχανημάτων είναι δυνατή και θα μπορούσε να είναι δυνατή ακόμα και η ανακύκλωση ε, στοιχείων, των κομματιών των μηχανημάτων αυτών. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να παραφ... θα πρέπει μάλλον να αναφτάσουμε σε μια αυστηρή εφαρμογή της ιεραρχίας των ε, ε διαφόρων αυτών ε, δράσεων για τα απόβλητα που έχουμε ήδη εγκρίνει. Θα ήθελα κάπως να με καθησυχάσετε και για αυτό που έλεγε ο συνάδελφος Παναγιώτοφ. Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα ε, περιέχουν στοιχεία που πολλές φορές είναι πολύ σπάνια και πολύτιμα. Και αν δεν καταφέρουμε να τα ανακτήσουμε, μπορεί να οδηγηθούμε σε μια ε, κατάσταση έλλειψης. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο συστηματικοί και συγκεκριμένοι για αυτή την υπόθεση. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα ήθελα να ξαναδούμε την οδηγία αυτή με βάση αυτές τις γραμμές, γιατί δεν θεωρώ πως είναι αρκετά ισχυρή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Λίζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υποστηρίζω τη θέση του Καρλ Χάιντς Φλόρεντς. Έχω μόνο τρεις ειδικέ παρατηρήσεις. Πρώτον, το θέμα των λαμπτήρων που εξοικονομούν ηλεκτρική ενέργεια. Πολλοί ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα και στον προεκλογικό αγώνα. Πολλοί θεωρούν ότι ο υδράργυρος δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν ισχύει αυτό το επιχείρημα γιατί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απελευθερώνεται ε, υδράργυρος. Συγγνώμη. Ε, ε στο ΓΟΥΙ όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται, αλλά εγώ δεν ξέρω κανέναν καταναλωτή που να πηγαίνει στο δημοτικό χώρο συλλογή για να πετάξει μία λάμπα ε, εξοικονόμηση ενέργειας. Βέβαια υπάρχει το επιχείρημα που λέει να έρχονται να το παίρνουν από το σπίτι σου, όπω προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά υπάρχουν και ενδιάμεσε λύσει. Το πιο απλό θα ήταν εκεί που αγοράζει αυτά τα πράγματα να μπορεί να τα επιστρέψει κιόλα. Θα ήταν πολύ πρακτικό έτσι, δεν είναι στις μπαταρίες, δεν το κάνουμε αυτό. Ε, και στο λιανικό εμπόριο και σε μεγάλες ε, αλυσίδες καταστημάτων γίνεται αυτό. Θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε, ε, μήπως να το κάνουμε κανόνα, να το γενικεύσουμε. Το δεύτερο, φωτοβολταϊκά. Εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία στους κατασκευαστές εγκαταστάσεων τέτοιων φωτοβολταϊκών συστημάτων ότι θα αυξηθεί πολύ το κόστος τους. Εδώ θεωρώ ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι λογική και δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε, να την ξεπεράσουμε. Και το τελευταίο για την αναδιατύπωση της οδηγίας. Έκκληση προς τον Πρόεδρο. Σωστά είπατε ως Πρόεδρος της Συνταγματικής Επιτροπής ότι το δικαίωμα πρωτοβουλίας έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά ήδη από την τωρινή διοργανική συμφωνία ορίζεται ότι σε περίπτωση που αυτό είναι σκόπιμο, if appropriate στα αγγλικά το λέει, ε, όταν ενδείκνυται μπορεί και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή να αλλάξει κάποια πράγματα χωρίς να το προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θέλω να απευθύνει ε, ενώ έκκληση να είμαστε πολύ γενναιόδοροι στην ερμηνεία αυτής της διάταξης για να είναι και πολιτική η έκθεση και να έχει και νόημα σε τελική ανάλυση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λίζε. Άμα το γράφει αυτό τότε θα το κάνουμε. Να δούμε και ποιες τροπολογίες θα κατατεθούν. Ο κύριος Σόνικ, παρακαλώ. Ε, θα, ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπαν ο Καρλ Χάιντ Φλόρενς και ο Ρίχαρτ Σίπερ. Την ανάγκη δηλαδή να δείξουμε πώς μπορεί να γίνει η συλλογή του ηλεκτρικού εξοπλισμού, για παράδειγμα στη χώρα μου, η παραγωγή δημιούργησαν ένα ταμείο, ένα ίδρυμα που αναλαμβάνει την συγκομιδή. Έχουν τοποθετήσει κάδους σε διάφορα σημεία. Υπάρχει όμως ε, αθέμητος ανταγωνισμός επιδρομής στους κάδους αυτούς και καταλήγει ο εξοπλισμός στη χωματερή όπου τα απόλυτα αυτά διατίθενται με τρόπο όχι πολύ φιλικό προς το περιβάλλον. Και τελικά δεν χρησιμοποιούνται οι σχετικές εγκαταστάσεις, διότι ο εξοπλισμός χάνεται κάπου σε κάποια γκρίζα ζώνη. Η οδηγία αυτή λοιπόν έχει οδηγήσει στην ύπαρξη νόμιμης αγοράς για την ε, συγκομιδή των αποβλήτων. Δεν υπάρχει όμως καμία εγγύηση ότι πράγματι ανακυκλώνεται σωστά ο εξοπλισμός αυτός. Νομίζω ότι αν μπορούμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτό με την αναδιατύπωση της οδηγίας, εάν μπορέσουμε αυτήν την εικονική αγορά να την κάνουμε πραγματική, Όσον αφορά δηλαδή την ανακύκλωση των επικίνδυνων ε, ουσιών, αυτό θα είναι χρήσιμο και για μας και για το περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ, ο Κρίστοφ Χέλνερ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ε, επαναλάβω αυτό που είπαν αρκετοί από τους προλαλήσαντες, ότι είναι περίεργο να επιλέγεται η αναδιατύπωση που περιορίζει τις δυνατότητές μας να ε, αναθεωρήσουμε αυτήν την πολύ συζητημένη οδηγία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε αν ενδείχνεται κάτι τέτοιο. Αλλά αυτά που προτείνονται γενικά τα βρίσκω καλά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πώς όλα αυτά επηρεάζουν το εμπόριο, ώστε να μην δυσκολεύεται το εμπόριο με τις νέες απαιτήσει και να γίνονται πιο πολύπλοκες οι διαδικασίες, διότι κάτι τέτοιες ανησυχίες ε, νιώθω όταν διαβάζω την πρόταση αυτή. Κάτι άλλο που μου λείπει είναι ότι νομίζω ότι έχουμε χάσει την ευκαιρία για αναρμόνιση με την ε, αναδιατύπωση, κάτι που ανέφερε και ο κύριος Ρίπερ και ο κύριος ε, ε Φλόρενς. Το θέμα είναι μάλλον οι διαφορές, στην εφαρμογή που θα οδηγήσουν σε δυσκολίες. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε τον βαθμό εναρμόνισης με την αναδιατύπωση. Και τέλος, υπάρχει ένας τομέας για τον οποίο δεν έχω πολλές γνώσεις, αλλά έχουμε εδώ μία οδηγία η οποία κυρίως ε, έχει να κάνει με τον οικιακό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Είναι όμως κάτι που επηρεάζει και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μεγάλες γεννήτριες για παράδειγμα. Θα πρέπει να φροντίσουμε να μην δημιουργήσουμε εδώ ένα σύστημα το οποίο να καλύπτει με διαφορετικούς τρόπους δύο ε, τελείως διαφορετικούς τομείς. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε, έναν βιομηχανι... σε, ανάμεσα σε μια βιομηχανική γεννήτρια και ε, στην ε, δική μου τηλεόραση. Αυτό θα πρέπει να το φροντίσουμε στην ε, νομοθεσία αυτή. Δύο λεπτά και 17 δευτερόλεπτα μίλησα. Δεν νομίζω ότι ξεπέρασα το χρόνο μου. Ναι, πράγματι, ο κύριος Ορέστε Ρώση, λέει ο πρόεδρος. Sì, grazie Presidente, sono d'accordo con quello che Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα όσα είπαν πολλοί συνάδελφοι. Πιστεύω πως είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η ανάκτηση των στοιχείων που βρίσκονται μέσα στις ηλεκτρονικές συσκευές και θα πρέπει να γίνεται αυτό συστηματικά ε, στα μεμονωμένα κράτη. Θα πρέπει να γίνεται η συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από πλευρά των παραγωγών. Γίνεται, ναι, μπορεί να γίνεται, αλλά πρέπει να υπάρχουν μια βασική προπόθεση ότι να υπάρχει δηλαδή υποχρέωση επιστροφής στους τους παραγωγούς. Να σα δώσω το παράδειγμα της Ιταλίας. Ένας πολιτή μπορεί να, να ξεφορτωθεί είτε το πλυντήριό του, είτε το τηλεόρασή του με διάφορα συστήματα. Είτε το πάμε στο, πάνε στο ε, στους ε, συλλέκτες ε, παλιών συσκευών που κάνουν την ανάκτηση αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πότε είτε στέλνουν στη, σε ειδικού οργανισμούς που στέλνουν τα παλιά, τις παλιές συσκευές στον τρίτο κόσμο για να τους βοηθήσουν. Λείπει λοιπόν η ενιαία συλλογή και πώς μπορούμε λοιπόν να αναθέσουμε ευθύνε στους ε, παραγωγούς χωρίς ε, με τη σειρά να υποχρεώνουμε και τον καταναλωτή να επιστρέψει στον παραγωγό το αντικείμενο της συσκευή και αυτό να γίνει και με πρόστιμα αν δεν ε, επιτευχθεί το συγκεκριμένο ποσοστό ανάκτησης αυτό το κόστος επιβαρύνει τον παραγωγό και φυσικά και αυτός με τη σειρά του θα επιβαρύνει τον χρήστη. Grazie, Karin Ευχαριστώ κυρία Κάντενπαχ. Ευχαριστώ. Μια διευκρινιστική ερώτηση. Όταν μιλάμε για 65% αναχώρα ή γενικώ και αορίστος. Γιατί μιλήσαμε για συμπεριφορές καταναλωτών. Ξέρουμε ότι στις μεγάλες συσκευές είναι πολύ μεγάλη η προθυμία να κάνουν απόσυρση. Στις μεγαλες συσκευέ ειναι συσκευές είναι πολύ μικρες συσκευέ Δηλαδή αυτό το ποσοστό τι παριστά. Μήπως ε, έχουμε πολύ μεγάλη στρέβλωση της συνολικής εικόνας όταν μιλάμε έτσι γενικά. Θα απαντήσει και ο κύριος Φλόρενς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σαμπίνεν Βίλτς. vielen Dank. Ähm, Ευχαριστώ πολύ. Καλό είναι να συνεχιστεί η οδηγία, να αναδιατυπωθεί για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που αποσύρονται και ε, καλωσορίζω την πρόταση καταρχήν, αλλά συμφωνώ και με την ερώτηση για το στόχο το 65%. Διάβασα ε, ότι ε, μπορεί να γίνει αυτό μετά από δύο χρόνια, όχι το 2016. Και κάτι άλλο που είναι ενοχλητικό ότι ο στόχος έχει να κάνει, λέει, με το βάρος της συσκευής και όχι με το είδος της συσκευή γιατί μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές συσκευέ μεταξύ τους. Και τελικά που μπορεί να οδηγηθούμε. μικρέ συσκευές, ελαφριές, MP3, να τις πετάνε στα σκουπίδια κανονικά και να αποσύρεις μια μεγάλη συσκευή και να φτάνεις στο στόχο του 65%. Αυτό πώς μπορούμε να το λύσουμε και να αποφύγουμε. Για να έχουμε και διαφορετική στάση ε, προς τα πράγματα και τις συσκευές. Η Φρανσουάζ Γκρουστέ, τελευταία, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ που με επιτρέπετε να παρέμβω. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Θέλω να επιμείνω για το πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας, ε, ζητώντας ε, να φροντίσουμε να αποκλειστούν τα φωτοβολταϊκά τόξα, γιατί ε, μέσα στο πλαίσιο της ε, καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών θέλουμε να προωθήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξέρουμε πως έχουμε μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί το, ένα στοιχείο του κάδμιου. Ε, είναι το λιγότερο δαπανηρό. αυτά τα... Οι ηλιακοί συλλέκτες είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι πιο φιλικοί στο περιβάλλον δεν παρουσιάζουν κίνδυνο οι ίδιοι για την υγεία ή για το περιβάλλον. Οι κατασκευαστές που παράγουν αυτά τα, τους φωτοβολταϊκούς συλλέκτες έχουν δεσμευθεί εθελοντικά σε συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης, δεδομένου ότι η διάρκεια ζωής τους είναι τουλάχιστον 25 χρόνια. Πιστεύω πως πρέπει άμεσα να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ε, τα φωτοβολταϊκά ε, αυτά οι συλλέκτες, γιατί διαφορετικά θα φρενάρουμε τη χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας. Ευχαριστώ. Το θέμα αυτό το άκουσαν οι αντίστοιχε εταιρείε την τελευταία εβδομάδα τι γίνεται με τους ηλιακούς συλλέκτες. Παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις πριν μας πει ο κύριος Φλόρεντς στη συνέχεια της διαδικασίας. Yeah, for... Ευχαριστώ πολύ που μας ξαναδίνετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τους σημαντικούς συλλογισμούς που μοιράστηκαν μαζί μας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφερθώ σε κάποιες από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν. Ε, καταρχήν, ο ρυθμός ε, συγκομιδής που προτείνουμε. Πράγματι, στις ε, πιο όριμες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη σήμερα. Ο βαθμός συγκομιδής πλησιάζει το 65% του εξοπλισμού που διαδέθηκε στην αγορά τα προηγούμενα χρόνια. Το ποσοστό συλλογής δηλαδή, ήδη δηλαδή ε, ε, πλησιάζουμε τον, το στόχο μας ε, και έτσι διαψεύδουμε αυτούς που λένε ότι είναι υπερβολικά φιλόδοξος ο στόχος αυτός ή δεν θα το πετύχουμε ποτέ. Ωστόσο, πρέπει να υποβάλουμε μια οδηγία που θα εφαρμόζεται στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη όπου το ποσοστό δεν θα είναι τόσο ψηλό, όπου δηλαδή διατίθεται ακόμα πολύ περισσότερος ηλεκτρονικός εξοπλισμός κάθε χρόνο από ό,τι συλλέγεται. Πιστεύουμε ότι με προθεσμία το 2016 θα έχουμε μια ημερομηνία όπου στα περισσότερα κράτη-μέλη θα έχουμε πετύχει το στόχο του 65%. Θα ήθελα ωστόσο να αναφέρω ότι στην πρόταση αυτή ε, δεν προχωράμε αδίστακτα. Έχουμε δύο δίκτυα ασφαλείας. Το 2012 σκοπεύουμε να επανέλθουμε με μια έκθεση σχετικά με τη σκοπιμότητα του, ε, με το κατά πόσο είναι επιτεύξιμος δηλαδή ο προτινόμενος στόχος. Η έκθεση αυτή μπορεί να εξετάσει και το θέμα της διαφοροποίησης. Το ακούσαμε αυτό και από κάποιους από εσά, γιατί δεν ε, εξετάσαμε διαφορετικές λύσεις για διάφορα είδη εξοπλισμού, τον ελαφρύ, τον μέτριο, τον πιο βαρύ, τον εξοπλισμό ψήξης, ε, θέρμανσης κλπ. Θα επανέλθουμε λοιπόν με έκθεση προς εσάς και ενδεχομένως θα υποβάλουμε σχετική πρόταση προσαρμογής του στόχου. Γιατί επιδιώκουμε το 85%? Φοβάμαι ότι μπορεί να μην εξαντλήσουμε το δυναμικό μας, αλλά πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να καλύψουμε τα διαθέσιμα απόβλητα, διότι υπάρχει κάποιο ποσοστό εξοπλισμού που παρά την ε, σχετική σήμανση τελικά καταλήγει στα κανονικά απορρίμματα. Το θέμα είναι λοιπόν να καλύψουμε και τα απορρίμματα αυτά. Θέλουμε δηλαδή να τα καλύψουμε και αυτά, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Αρχικά θέλαμε να καλύψουμε το 87%, τώρα θέλουμε να καλύψουμε το 85%. Θα πρέπει όλα αυτά τα απόβλητα να διατίθεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας. Για να διασφαλίσουμε κάτι τέτοιο, ζητήσαμε πλήρες καθεστώς λογοδότησης. Θέλουμε δηλαδή τα κράτη-μέλη στο τέλος της χρονιάς να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με το 85%. όσον αφορά τους στόχους και την ανακύκλωση ανακατηγορία. Θα βρείτε αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις διάφορες κατηγορίες. Θεωρήσαμε ότι η διαφοροποίηση των στόχων θα μας οδηγούσε σε μια υπερβολικά πολύπλοκη κατάσταση όπου και οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων θα ήταν υπερβολική. Και θα επαναρχόμασταν έτσι σε διοικητικό φόρτο ανάλογα με αυτόν από τον οποίο προσπαθούμε να ξεφύγουμε. Ελπίζω να απάντησα στις βασικές ανησυχίες που εκφράστηκαν. Ευχαριστώ που μας δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ο Καλχάιντς Φλόρενς. Πώς θα προχωρήσουμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι άκουσα πολλά, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ακούσαμε κάποιες φωνές υπέρ της εναρμόνισης. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν γιατί το Συμβούλιο επιμένει με πολύ πείσμα στις εθνικές ρυθμίσεις των τομέα αυτών τη στιγμή που συμφωνούν και τα 27 κράτη-μέλη. Η καταχώρηση στα διάφορα κράτη-μέλη αποτελεί πηγή εισοδήματος ε, για τις κυβερνήσεις. Ίσως γι' αυτό επιμένουν τόσο πολύ στο να διατηρήσουν τα συστήματά τους. σε ε, αναπτυσσόμενες χώρες ε, δεν μπορεί να συλλέξει κανείς ε, τον εξοπλισμό που έχει πολιθεί τα δύο τελευταία χρόνια για ευνόητους λόγους. Οπότε η σύγκριση αυτή δεν είναι πολύ σωστή, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε διμέρως με την Κομισιόν. κύριε Πρόντι ευχαριστώ πολύ για την σχετική ιεραρχία. Δεν θα πρέπει όμως να καταλήξουμε σε ένα τόσο πολύπλοκο σύστημα που να απαιτούμε πανάρχια ψυγεία όπως το ψυγείο της μητέρας μου, που ήταν 28 ετών, να ανακυκλωθεί. Καταπίνουν τόσο πολύ ενέργεια αυτά τα αυτές οι συσκευές που δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε. Η Κομισιόν προτείνει ποσόστοση 85% συλλογής και ανακύκλωσης. Ε, μπορεί να το συζητήσει κανείς αυτό, κύριε Ρώση. Δεν κατάλαβα τη χθεσινή σας παρέμβαση, αλλά και τη σημερινή σας δεν την κατάλαβα καθόλου. Πείτε μου τι ακριβώς θέλετε. Στην Ιταλία έχουμε χειρότερες ποσοστώσεις ε, συγκομιδής από ό,τι στη Βουλγαρία. Και αυτό... Και γι' αυτό δεν, δεν ε, ευθύνονται οι πολίτες της Ιταλίας, η ρύθμιση ευθύνεται. Πιστέψτε με, θα πρέπει να πάρετε θέση, θα πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα στην Ιταλία ότι θέλετε να συλλέξετε τον εξοπλισμό και οι πολίτες θα φέρουν τα παλιά τους, τις παλιές τους συσκευές. Ε, θα χαρώ πολύ και με οποιαδήποτε παρατήρηση λάβω σε διμερές επίπεδο. Να σας πω ότι όσον αφορά την προθεσμία έχω κάποιες επιφυλάξεις. Θα προσπαθήσω. Αλλά δεν μπορώ να τους υποσχεθώ ότι θα τηρήσουμε όλες τις προθεσμίες και για την ε, παράλληλη ρύθμιση ΡΟΣ. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια. Παρακαλώ όμως να δείξετε κατανόηση εάν δεν προλάβουμε τις προθεσμίες. Μπορεί να υπάρχουν πολύ λίγε μέρες ανάμεσα στην υποβολή τη εκθεσή μου και την προθεσμία για τις τροπολογίες. Ε, αυτό θα οφείλεται στο γεγονό ότι θα θέλω να τηρήσω τι προθεσμίες, θα κάνω ό,τι μπορώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Απαντήσατε ε, στον κύριο Ρώση. Νομίζω θα θέλει να σα εξηγήσει τι ακριβώ είπε. Σύντομα, κύριε Ρώση. Ε, Συνήθω δεν το κάνουμε, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση θα, θα ακούσουμε τι έχετε να πείτε. Ε, Όχι, είναι απαραίτητο, Προέδρε, γιατί δεν ε, συνονοηθήκαμε. Δεν είπα τίποτα από αυτά που αναφέρθηκαν. Εγώ είμαι υπέρ στην ανάκτηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Αλλά ανέφερα ένα πρόβλημα για την Ιταλία, για παράδειγμα, όπου σήμερα αυτέ οι συσκευέ μπορούν να ανακτηθούν με τρει τρόπου. Ένα, μέσω τη συλλογή που κάνουν οι τοπικέ αρχέ, δηλαδή δήμοι. Δεύτερον, μέσω τη συλλογή που κάνουν κάνουν ε, ιδιώτες ε, συλλέκτες και μετά τα ανακτούν δεν ξέρω ακριβώς πώς, είτε μέσω εθελοντικών συνδέσμων που συλλέγουν και στέλνουν μετά τα συσκευέ που ακόμα λειτουργούν σε τρίτες χώρες ως βοήθεια. Αν εμείς θέλουμε να αναθέσουμε ευθύνες στους παραγωγούς, για την ανάκτηση θα πρέπει να καταστήσουμε την ανάκτηση υποχρεωτική και μάλλον την επιστροφή υποχρεωτική και για τον καταναλωτή. Δεν γίνεται διαφορετικά να επιβάλλουμε πρόστιμα στους παραγωγούς μόνο επειδή δεν κατάφεραν να φτάσουν σε συγκεκριμένο ποσοστό ανάκτησης γιατί ούτως ή άλλως το κόστος αυτό θα έχει αντίκτυπο και στους καταναλωτές. Ωραία. Ο κύριος Φλόνες κατάλαβε τώρα τι θέλετε να πείτε. Ωραία. Και έχουμε και την ερώτηση προς το Συμβούλιο γιατί αντιστέκεται στην εναρμόνιση. Θέλετε να παρέμβετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Από την πλευρά της Προεδρίας, λίγα λόγια από τη δουλειά που γίνεται στο Συμβούλιο πάνω στο συγκεκριμένο νομοθέτημα. Ο στόχος της απλοποίησης και τη συγκομιδής και ανάκτησης των προϊόντων αυτών. Είναι στόχος που συμμερίζονται τα δύο θεσμικά όργανα που ασχολούνται με την αναδιατύπωση της ε, οδηγίας. Λίγο πολύ όλα τα κράτη-μέλη συμφωνούν ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να πετύχουμε την απλοποίηση αλλά να διασφαλίσουμε παράλληλα ασφαλή προς το περιβάλλον εφαρμογή της νομοθεσίας, για την νομοθεσία αυτή που εφαρμόζεται για σχετικά βραχή χρονικό διάστημα θα ήταν να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με βάση τα εθνικά συστήματα, ωστόσο με σημαντικές βελτιώσεις ως προς τον τρόπο εφαρμογής, δηλαδή να υπάρχει απλοποίηση για τους διάφορους παράγοντες και τους καταναλωτές και τους παραγωγούς και τους άλλους φορείς που συμμετέχουν στην εφαρμογή της οδηγίας για να διασφαλιστεί η σωστή και φιλική προς το περιβάλλον εφαρμογή της οδηγίας. Ε, προσβλέπουμε στις ε, συνομιλίες ε, με τον εισηγητή και άλλους ενδιαφερομένους πάνω στο θέμα αυτό. Και κλείνοντας, ε, να σας ενημερώσω ότι κατά τη διάρκεια της προεδρίας αυτής ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω στο θέμα αυτό. Είχαμε μια συζήτηση πολιτικής, μια πολιτική συζήτηση όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας και θα διασφαλίσουμε την ομαλή μετάβαση ε, στην επόμενη προεδρία όσον αφορά το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ. Από πλευρά μεθόδου και χρονοδιαγράμματος, καλό θα ήταν να το έχουμε και τα δύο αυτά παράλληλα στην Ολομέλεια. Περίπου ταυτόχρονα, για να μην πω ακριβώς ταυτόχρονα, να έχουμε και την ε, ψηφοφορία και τις εκθέσεις. Τέλη λοιπόν Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου σχέδιο έκθεσης. Τον Απρίλιο ψηφοφορία στην Επιτροπή και το Μάιο από ό,τι φαίνεται στην Ολομέλεια. Έτσι είναι ο σχεδιασμός. Και τώρα ερχόμαστε στο επόμενο ζήτημα, στο 12. Περιορισμοί στη χρήση ε, ορισμένων επικινδύνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ε, η συγγήτρια είναι η κυρία Jill Evans. Θα ήθελα να της δώσω το λόγο για να μας κάνετε μια εισαγωγή παρακαλώ στο θέμα. Ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω πως η Κομισιόν ήθελε καταρχήν να παρουσιάσει το θέμα και μετά να σας πω και εγώ τις ιδέες μου για την ε, έκθεση. Α, το θέλετε αντίστροφα. Καλά. Η Κομισιόν πρώτα να μας πει τι προτείνει. Ο κύριος Κιούκλερ. Yeah, thank um, can... Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω πως ε, θα σας εξηγήσω την... τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της πρότασης σχετικά σύντομα. Για ποιο λόγο προτείνουμε και ποια ήταν, ποιο ήταν το σημείο κίνησής μας. Καταρχήν, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, όπου αρχίσαμε να κοιτάμε να εξετάζουμε μάλλον την αναθεώρηση, είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπου έχουμε ένα νέο είδος νομοθεσίας ε, που βασικά μόλις άρχιζε να λειτουργεί και να γίνεται γνωστό και κατανοητό από τους ε, ενδιαφερόμενους φορείς. Ωστόσο μπορούσαμε ήδη να δούμε ότι οι πρώτες εμπειρίες έδειχναν, όπως και με την οδηγία αυτή, κάποιες αδυναμίες στην εφαρμογή, κάποια προβλήματα εφαρμογής και συνοχής ε, ανάμεσα στα κρατημέλη, πράγμα το οποίο προκαλούσε περιττό διοικητικό φόρτο και νομικές επιπλοκές. Επιπλέον η οδηγία ζητούσε από την Κομισιόν να εξετάσει κάποιες πτυχές, δηλαδή την συμπερίληψη των κατηγοριών 8 και 9, δηλαδή ηλεκτρικές συσκευές και συσκευές μέτρησης και να δούμε επίσης τον κατάλογο με τις επικίνδυνες ουσίες για να τον τροποποιήσουμε αναλόγως. Εμεί προβήκαμε στην αναθεώρηση με, τον ακριβώς, με ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως κάναμε και στην WE. Θεωρήσαμε πως ήταν σωστό λόγω της, του μικρού χρονικού διαστήματος ισχύω της ε, νομοθεσία να μην κάνουμε κάποια επαναστατική αλλαγή, να ξεφορτωθούμε τα πάντα και να επανέλθουμε με κάτι τελείω νέο, αλλά να εξελιχθούμε και να κάνουμε μια εξελιχτική πρόταση ώστε να βελτιώσουμε αυτά που προφανώς δεν λειτουργούσαν. Γι' αυτό και θεωρήσαμε πως μια πρόταση αναθεώρησης θα ήταν πιο σωστή σε μια τέτοια περίπτωση. Να σας πω λοιπόν ποια είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης. Δεν αγγίξαμε τους βασικούς στόχους βεβαίως. Οι βασικοί στόχοι είναι να εξαλειφθούν κάποιες επικίνδυνες ουσίες από τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές και αυτό με στόχο να προστατευθούν όλοι όσοι εργάζονται με αυτές τις συσκευές από τη στιγμή που αυτές είναι πια απόβλητα και Φυσικά να προστατεύσουμε και το περιβάλλον από την απελευθέρωση αυτών των ουσιών όταν θα μπουν στη διαδικασία κατεργασίας αποβλήτων. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι καθορίζεται από τη δυνατότητα να εξερεχθούν κάποιες τεχνικές εφαρμογές από την απαγόρευση όταν και αν μια τέτοια προσωρινή εξαίρεση θεωρηθεί απαραίτητη επί τεχνολογικής ε, βάσης, δηλαδή αν δεν υπάρχουν υποκατάστατα. Και προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε το στόχο αυτό ε, ως είχε. Η πρώτη μεγάλη αλλαγή που προτείναμε, τη συζητήσαμε, δεν χρειάζεται να επανέλθουμε σε αυτήν με όλε τι λεπτομέρειε, ήταν να αντιστρέψουμε τη σχέση ανάμεσα στι δύο οδηγίε. Στην πρότασή μας αυτή η οδηγία είναι η οποία προηγείται και η οδηγία WE είναι αυτή που δίνει, ε, που ακολουθεί Έχουμε διευκρινίσει διάφορους ορισμούς που προκάλεσαν μεγάλες αβεβαιότητες και τους έχουμε ευθυγραμμίσει με νεότερες νομοθεσίες που έχουν προκύψει όπως για παράδειγμα την έννοια του οικονομικού φορέα. Επίσης, τι είναι οι ιατρικές συσκευές και έχουμε επίσης ενσωματώσει την έννοια των ομογενοποιημένων υλικών. Ένα από τα πιο δύσκολα σημεία ήταν το θέμα της τροποποίησης ε, της απαγόρευσης ουσιών. Για αυτό το θέμα προχωρήσαμε ως εξής. Κάναμε μια πολύ μεγάλη διερεύνηση των πιθανών ουσιών που χρησιμοποιούνται και που για κάποιο λόγο ανέπιπταν στο πεδίο και ελέγξαμε αυτές τις ουσίες για να δούμε αν υπάρχουν αποδείξεις για το αν και πώς θα έπρεπε και πότε θα έπρεπε να προσθεθούν στον κατάλογο. Νομίζω πως αυτό η υπόθεση είναι γνωστή. Από ένα πολύ μακρύ κατάλογο τελικά καταλήξαμε σε πέντε σοβαρούς υποψήφιους τελικά Και έπειτα όταν ελέγξαμε προσεκτικά αυτούς τους πέντε σοβαρούς υποψηφίους, διαφοροποίησαμε ανάμεσα σε έναν και αυτή η ουσία λέγεται TBBBA. Είναι ένα υλικό κατά της ανάφλεξης Πιστεύαμε ωστόσο πως ε, η ήδη υπάρχουσα στρατηγική ήταν επαρκής και δεν χρειαζόταν να υπάρξει διπλή νομοθεσία προ αυτό. Ε, οι υπόλοιπε τέσσερις ουσίε και δεν θα σα αναφέρω τα το ονόματά τους, εντοπίστηκαν... Ήταν ε, ουσίε για τις οποίες δεν είχαμε και γι' αυτό δεν τις προσθέσαμε στον κατάλογο, δεν είχαμε σε αυτή την χρονική στιγμή επαρκή πληροφορίες πρώτον για την ε, διαθεσιμότητα υποκατάστατων που είναι πολύ σημαντική, αλλά ούτε και για το κόστος ωφέλεια. Τη σχέση μάλλον κόστος ωφέλεια εν μια πιθανή απαγόρευση. Άρα λοιπόν αποφασίσαμε ότι θα ήταν καλό να εντοπίσουμε με αυτές τις τέσσερις ουσίες ως ε, τις ε, πιο πιθανές υποψήφιες για μελλοντική απαγόρευση, αλλά ότι θα έπρεπε να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες πριν αποφασίσουμε για κάτι τέτοιο. Πέρα από την απαγόρευση των ουσιών, και αυτό είναι ίσω το δεύτερο σημαντικότερο θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί, είναι το πώς θα γίνει ο εντοπισμός των ουσιών που πρέπει να απαγορευθούν στο μέλλον. Και μετά να προτείνουμε μια ευθυγραμμισμένη προσέγγιση όσο αυτό είναι εφικτό και λογικό με τη νέα χημική νομοθεσία που έχει εντωμεταξύ υιοθετηθεί, από, δηλαδή το REACH. Και γι' αυτό Και γι' αυτό είπαμε ότι και μια μελλοντική διαδικασία Ρώσ για την απαγόρευση ουσιών θα πρέπει να ακολουθεί και τη βάση ε, τις βάσεις του ΡΙΤΣ, αλλά δεν θα πρέπει να εμπίπτει μέσα στη λήψη αποφάσεων του ΡΙΤΣ. Το ΡΟΣ δηλαδή θα πρέπει να έχει τη δική του ζωή, αν και από επιστημονικής άποψης θα, θα ακολουθεί την προσέγγιση του ΡΙΤΣ. Μετά είδαμε το δεύτερο στοιχείο, είπαμε είναι η απαγόρευση των ουσιών, προσωρινές εξαιρέσεις, εδώ έχουμε εισάγει δύο νέα στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι αντιστερέφεται το βάρος απόδειξης. Από εδώ και μπρος θα είναι απαραίτητο εκείνοι που θέλουν να πετύχουν μια ανεξαίρεση να αποδείξουν και να δώσουν τις αποδείξεις πως όντως τιολογείται μια εξαίρεση. Ενώ αυτή τη στιγμή το βάρος της απόδειξης ε, ανήκει στην Κομισιόν και κάποιες φορές ε, αυτό το καθήκον ε, είναι οριακά εφικτό. Και επίσης αυτό συμφωνεί με το ΡΙΤΣ και άρα οδηγεί σε μεγαλύτερη εναρμόνιση ανάμεσα στις διάφορες νομοθεσίες. Αξίσου προτείναμε την εισαγωγή ή μάλλον ε, την καλύτερη αιτιολόγηση ε, χορήγησης εξαιρέσεων ε, και αυτό επί τη βάση του ότι σήμερα βρισκόμαστε σε διαφορετική κατάσταση από ότι ε, πριν από 7-8 χρόνια. Γιατί σήμερα έχουμε όλοι συμφωνήσει σε πολλές νομοθεσίες και σε ευρωπαϊκές στρατηγικές ότι η βιώσιμη ανάπτυξη βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Πυλώνας ε, πρώτος είναι το περιβάλλον, αλλά επίσης κοινωνικο-οικονομικοί πυλώνες. Και Γι' αυτό και πιστεύουμε πως είναι δίκαιο και σωστό να χρησιμοποιούνται και οι τρεις πυλώνες αυτοί όταν εξετάζουμε αίτια για την χορήγηση εξαιρέσεων. Λόγος μάλλον για τη χορήγηση εξαιρέσεων. Ξέρουμε ότι όντω η υποκατάσταση ουσιών καταρχήν είναι δυνατή σε πολλέ περιπτώσει, αλλά για παράδειγμα κανεί σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να παρέχει στην αγορά τι απαραίτητε ποσότητε. Αν παρόλα αυτά απαγορεύσουμε μια εφαρμογή υπό τέτοιε συνθήκες, μπορεί σοβαρά να ζημιώσουμε ε, την θέση απασχόληση στην Ευρώπη. Γι' αυτό και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης. Η οδηγία πάσχει από ατελή εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Με την έννοια ότι η εποπτεία της αγοράς δεν είναι αρκετά αυστηρή. Και αυτό σημαίνει ότι διάφοροι μοναχικοί καβαλάριδες ξεφεύγουν πολύ εύκολα. Και γι' αυτό και έχουμε βάλει και στα άρθρα 6 με 8 νέους μηχανισμούς ώστε να αποδεικνύουμε την συμμόρφωση των προϊόντων και έχουμε προτείνει εδώ ότι με περισσότερες λεπτομέρειες από ό,τι θα μπορούσαν να υπάρχουν στο μέλλον μέσα στο πλαίσιο της ε, διαδικασίας επιτροπολογίας. Να ολοκληρώσω λέγοντας σύντομα τι δεν έχει γίνει, γιατί προφανώς παρακολουθούμε διάφορες επιλογές που στο τέλος μιας αξιολόγησης έχουμε ίσως παραβλέψει για διάφορους λόγους. Σίγουρα δεν έχουμε ακολουθήσει εκείνε τις φωνές που πρότειναν την γενική εκβάθρον αναθεώρηση τη οδηγία για πολλούς βάσιμους λόγους, γιατί πιστεύουμε πως ε, έχει λόγο ύπαρξης εκτός, ε, ε, παράλληλα με την νομοθεσία για τα χημικά. Δεν ακολουθήσαμε την τις που έλεγαν να αναθεωρηθεί απαγόρευση για το δεκαμπίλ. πιστεύουμε ότι θα πρέπει να παραμείνει απαγορευμένο. Προφανώς δεν επιλέξαμε και την επιλογή του να μην κάνουμε τίποτα. Και για την ώρα δεν προτείνουμε την αναθεώρηση του καταλόγου απαγορευμένων ουσιών λόγω της ε, ε αβεβαιότητας των στοιχείων. Προτείνουμε ωστόσο να εξετάσουμε επιγόντως όλες αυτές τις ουσίες. Αυτά συναπτικά το περιεχόμενο της πρότασής μας. Ευχαριστώ. Euh. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στη Jill Evans, αν θέλει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Κούγκλερ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη τόσο σαφή παρουσίαση της αναδιατύπωσης ε, των περιορισμών ε, επικινδύνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Καταρχήν πρέπει να πω ότι συμφωνώ με πολλά από τα σημεία που μας ανέφερε. Στόχος της οδηγίας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και η συνεισφορά ε, στην απόσυρση ε, με τρόπο αηφόρο. Δηλαδή το θέμα δεν είναι μόνο η απόσυρση των αποβλήτων και η διαχείριση των αποβλήτων, αλλά η πιο πράσινη οικονομία όπως είπαμε προηγουμένως, ε, τα περισσότερα απόβλητα παράγονται από ε, αυτά τα προϊόντα. Μιλάμε για 9 εκατομμύρια τόνους ετησίως και μέχρι το 2020 θα έχουν γίνει 12 εκατομμύρια τόνοι ετησίως αυτά τα απόβλητα. Και ε, συνήθως φεύγουν ουσίες, διαφεύγουν ουσίες χωρίς να το θέλουμε στο περιβάλλον και πολλές φορές έχουμε και λαθρές εξαγωγές σε τρίτες χώρες ε, αναπτυσσόμενες με πολύ σοβαρά προβλήματα διότι κατά τη διάρκεια ε, της μετατροπής τους ε, γίνονται διοξίνες ας πούμε οι ουσίες αυτές. Υπάρχουν βαρέα μέταλλα και ουσίες επιβράδυνσης της φλόγας για ασφάλεια αλλά ε, και όλες οι ρυθμίσεις δεν ε, ήταν ε, απαγορευτικές. Πολλές εταιρείες προχώρησαν σε νέα τεχνολογία και πολλές μάλιστα δεν χρησιμοποιούν καν βρωμιούχες ή χλωριούχες ουσίες πλέον. Είναι λοιπόν καλή η προσπάθεια που κάνετε, να βήμα πιο πέρα και... καλή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να σας αναφέρω τάχει κάποια σημεία στα οποία θα εστιαστεί και το δικό μου έγγραφο. Για το πεδίο εφαρμογή έγινε πολλής λόγος ποια προϊόντα θα πρέπει να καλύπτει η οδηγία αυτή. Και το επιχείρημα ήταν να υπάρχει ένας κατάλογος δεσμευτικός για καλύτερη εναρμόνιση και λιγότερη σύγχυση για το τι εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογή και τι όχι. Αλλά ο δεσμευτικό κατάλογο δεν μπορεί να καλύψει ε, τη ταχύτητα με την οποία αναπτύσσονται και κυκλοφορούν νέα προϊόντα. Δεν είναι λοιπόν ε, εξαντλητικός και δεσμευτικός ο κατάλογος γιατί αναφέρει τους, τις κατηγορίες στις οποίες θα χωρίζονται τα προϊόντα. Δεν είναι λοιπόν δεσμευτικό, ε, ούτε καλύπτει τα πάντα ο κατάλογο αυτό. Πιστεύω λοιπόν μόνο ότι ένα ανοιχτό πεδίο εφαρμογή θα λύσει το πρόβλημα των διαφόρων ερμηνεών. Δηλαδή καλύπτουμε όλα όσα δεν ξερούνται από το πεδίο εφαρμογής. Αυτό θα βελτιώσει την νομική βεβαιότητα και πιστεύω ότι στο Συμβούλιο υπάρχει ευρεία υποστήριξη για το θέμα αυτό. Αυτό λοιπόν προτείνω. Μαζί με αυτό όμως ε, προτείνουμε και μια μεταβατική περίοδο για όλα τα προϊόντα που δεν καλύπτονταν πριν με την ίδια δυνατότητα εξαίρεση που θα αποτελέσει αντικείμενο συναπόφαση. Το δεύτερο θέμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι αυτό των νέων περιορισμών. Η οδηγία ΡΟΣ οδήγησε σε προϊόντα πυλαγμένα από μόλιβδο και κάδμιο. Έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε. Πιστεύω ότι και άλλες και άλλες ουσίες θα πρέπει να περιοριστούν. Θα πρέπει να γίνει η προσαρμογή του καταλόγου με βάση τις πρόοδου της επιστήμης. Αυτός ήταν ο στόχος αυτής ε, της ε, αναθεώρησης. Η μελέτη ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης, η οποία επίσης συστήνει περαιτέρω περιορισμούς. Η έκθεσή μου λοιπόν θα προτείνει κανόνες που να ακολουθούν αυτές, ε, αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, στο παράθυμα 3 είχαμε ουσίες που είχαν επιλεγεί για να αποτελέσουν αντικείμενο αναθεώρησης ε, και μπορούν να μεταφερθούν στο ε, παράθυμα 4. Θα εξετάσουμε και άλλες ουσίες με στόχο την σταδιακή κατάργηση κάποιων ουσιών όπως είναι το PVC. τις ε, αντιπυρικές ουσίες ε, και το PVC ε, ε, τις καταργούμε σταδιακά σε, σε, για χρήση σε κινητά τηλέφωνα και σε υπο, υπολογιστές. Οι εταιρείες όπως η Apple και η Sony Ericsson θα συζητήσουν τις δικές τους εμπειρίες σε μια διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί εδώ στο Κοινοβούλιο 18 Νοεμβρίου μαζί με την Κέμσεκ. Θα εξετάσουν πώς οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μετακινούνται από την χρήση επικίνδυνων ουσιών στις βιώσιμες λύσεις. Ήδη υπάρχουν φορείς, για παράδειγμα, που απονείμουν που δίνουν εγκρίσεις σε προϊόντα που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Αυτό δείχνει ότι οι αλλαγές που προτείνω δεν είναι μόνο δυνατές, είναι και πρακτικές. Κάποιες πρωτοβουλίες ε, είναι ευπρόσδεκτες, δεν αρκούν όμως. Θα πρέπει όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να συμμετέχουν ε, συμπεριλαμβανομένων των εταιριών που ε, κατασκευάζουν συσκευές οικιακού εξοπλισμού. Για να αποφύγουμε τις παρεξηγήσεις προτείνω οι, νέες, νέοι περιορισμοί για τις ουσίες αυτές να εφαρμόζονται στα καταναλωτικά προϊόντα, όχι στις ε, φαρμακευτικές ε, συσκευές ε, και λοιπά. Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά προϊόντα. Κάποιοι είπαν ότι θέλουν ε, να γίνεται ανάκτηση των ε, ηλεκτρονικών συσκευών μόνο ε, σύμφωνα με, την, το REACH. Αυτό όμως δεν με βρίσκει σύμφωνη. Η οδηγία ΡΟΣ ασχολείται με θέματα αποβλήτων που δεν κάνει η οδηγία ΡΟΣ. Η οδηγία, Ρίτς. Η οδηγία λοιπόν θα πρέπει να συμπληρώνει την ΡΙΤΣ για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις. Η λογική συνέπεια όλων αυτών είναι ότι για την οδηγία ΡΟΣ θα πρέπει να αναπτυχθούν ξεχωριστά κριτήρια και μεθοδολογία. Η οδηγία αυτή υιοθετήθηκε με τη διαδικασία της συναπόφασης και η πιο βασική λειτουργία της οδηγίας αυτής, η απόφαση δηλαδή σχετικά με τον περιορισμό των ε, επικίνδυνων ουσιών, θα πρέπει να ε, αποτελεί επίσης αντικείμενο συναπόφασης και όχι να αφαιθεί στην επιτροπολογία όπως προτάθηκε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να διατηρήσει το Κοινοβούλιο εδώ τις αρμοδιότητές του, καθότι η μεθοδολογία στην πρόταση της Επιτροπής δεν ορίζεται σαφώς. Θα πρέπει να συμμετέχουμε στην ε, θεμελιώδη διαδικασία του να αποφασίσουμε ποιες και πώς ε, θα περιορίζονται οι νέες, ποιες ουσίες θα περιορίζονται και πώς. Όσον αφορά τις εξαιρέσεις, θα Ήθελα να διατηρήσουμε το παρόν σύστημα με κάποιες τροποποιήσεις όμως. Ε, συμφωνώ απόλυτα με την απόφαση της ε, Επιτροπής ε, να αντιστρέψει το βάρος της απόδειξης από τους αυτούς τους στην στη βιομηχανία. Θα πρέπει δηλαδή η βιομηχανία να ζητά εξαίρεση. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα πρέπει να θέσουμε προθεσμία για την Κομισιόν έξι μήνες πριν την λήξη μιας παρέκκλησης που είναι χρόνος επαρκής για την Κομισιόν για να λάβει νέα απόφαση. Υπήρχαν κάποιες ανησυχίες σχετικά με την αβεβαιότητα για τις προθεσμίες ε, της βιομηχανίας. Πιστεύω ότι έτσι μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν πιστεύω ότι η ανεπάρκεια υποκατάστατων θα πρέπει να αποτελέσει λόγο να παρασχεθεί τετραετής παρέκκληση. Πιστεύω ότι μετά τη λήξη μιας παρέκκλησης θα πρέπει να υπάρχει μια περίοδος χάριτος, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να εξετάσουν ε, τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις. Η παρέκκληση δηλαδή δεν χρειάζεται να ανανεώνεται για τετραετία. Και τα κοινωνικο-οικονομικά θέματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε αυτά τα πλαίσια. Επίσης, ε, η Πιστεύω ότι η πρότασή μου θα ενθαρρύνει την πρόοδο όσον αφορά την εξέβριση εναλλακτικών λύσεων. Η Κομισιόν ε, κατανοεί και σέβεται τους κανόνες αυτούς. Θέλουμε να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτό για να διασφαλίσουμε την ε, μέγιστη προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Περιμένω να ακούσω τις παρατηρήσεις των σκιωδών εισηγητών και να σας θυμίσω για άλλη μια φορά ότι στις, Νοεμβρίου, στις 18 Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσουμε διάσκεψη όπου θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με κάποιους ε, από τους βασικούς παράγοντες της ε, βιομηχανίας pour trois minutes, si chaque intervenant veut bien prendre Σας ευχαριστώ κύριε Σονίκη. Τρία λεπτά, κάθε ομιλητής τρία λεπτά μπορεί να έχει. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με την γνώμη που ακούστηκε ότι δηλαδή θα πρέπει να σχετίζεται οπωσδήποτε με το ρίτς, ότι θα πρέπει η ΡΟΣ να είναι εναρμονισμένη. και ότι θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις μόνο εφόσον έχουν ζητηθεί. Η διάρκεια τώρα μιας εξαίρεσης είναι χωρίς διάρκεια η χορήγηση της εξαίρεσης. Πιστεύω πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να είναι δυνατόν. Θα πρέπει να σκεφτούμε ίσως τα τέσσερα χρόνια είναι πολύ λίγα ε, όσον αφορά τις νέες ουσίες και τα υποκατάστατα. Ίσως θα έπρεπε να δούμε τα διάφορα προϊόντα, διαφορετικά προϊόντα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ως υποκατάστατα. Για ορισμένες συσκευές ίσως θα χρειαζόταν ε, μακρύτερη χρονική περίοδος. Σημαίνει βέβαια αυτό και τεχνολογική διαδικασία πιο μακρά. Ε, ίσως να πρέπει να προβλεφθούν και εκεί εξαιρέσεις. Πιστεύω πως στις 18 πρέπει να εξετάσουμε όλα αυτά τα θέματα για να μπορέσουμε σύντομα να κλείσουμε τις εργασίες από αυτές τις οδηγίες. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Chris Davis. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. 85% των ηλεκτρικών, ηλεκτρικών αποβλήτων στην Ευρώπη συλλέγονται και είναι εντυπωσιακό το πόσο δεν ανακυκλώνονται και τελικά καταλήγουν ε, στους στοχούς και τα παιδιά της Αφρικής, της Ινδίας και της Κίνας καταλήγουν στο να δηλητηριάζουν εκείνους τους ανθρώπους και να χαλούν το δικό τους περιβάλλον. Πρέπει λοιπόν να χειριστούμε και το θέμα των παράνομων αποβλήτων και αυτή η οδηγία που καθιστά τα προϊόντα πιο ασφαλή τα ίδια σίγουρα θα βοηθήσει στο να μειωθεί το πρόβλημα. Πρέπει να είδα γύρω στους 30 εκπροσώπους των διαφόρων ομάδων πίεση την τελευταία εβδομάδα. Με λίγες εξαιρέσεις τους αρέσει η αρχή του ΡΟΣ. Ε, και τους αρέσουν οι προτάσεις που κάνει η Κομισιόν. Θέλουν μεγαλύτερη βεβαιότητα για το νόημα ορισμένων απαιτήσεων της οδηγίας, θέλουν μεγαλύτερη συνοχή στην εφαρμογή. Τονίζουν τα κράτη-μέλη ότι ερμηνεύουν ε, τους κανόνες με διαφορετικούς τρόπους και ότι πολύ συχνά η μεγάλη παραγωγή, η Χιούλε, η Πάκαρντ και οι τέτοιοι της ηλεκτρονικής βιομηχανία που έχουν ε, ηγηθεί στην εφαρμογή του ΡΟΣ επειδή φοβούνται ότι μπορεί να τους βουτήξουν σε κάποια χώρα ε, αντί να πιεστούν να το κάνουν αυτό από τις ε, νομικές ρυθμιστικές αρχές της χώρας το κάνουν από μόνοι Άρα λοιπόν η νομοθεσία προωθεί την καινοτομία και την, την κατάσταση. Ίσως θα έπρεπε να υποστηρίξουμε και την αρχή της ανοιχτής, του ανοιχτού πεδίου. Ένα, ε, γι' αυτό και αναφέρεται και αυτό το πάνελ. Επίσης είναι ενδιαφέρον, μια από τις επικρίσεις είναι η έλλειψη συνέπειας ή εναρμόνισης με τις προτάσεις REACH. Εγώ μίλησα ήδη κατηδίαν χτε με τον ε, Διευθυντή τη Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, όταν ήταν εδώ. Μου είπε ότι βεβαίω η νομοθεσία πρέπει να βελτιωθεί, αλλά το ΡΟΣ υπάρχει και λειτουργεί. Ενώ το ΡΙΤΣ δεν θα είναι εφαρμοστέο σε όλα τα προϊόντα για 5-10 χρόνια. Οπότε Ας μην το κάνουμε λάθος, ε, θα μπορούσαμε να το ξαναδούμε όταν θα ε, αναθεωρηθεί εκ νέου. Αλλά για την ώρα είπε συνεχίστε με το ΡΟΣ. Αφού αυτό το λέει αυτό λοιπόν, ε, νομίζω ότι δεν υποτίθεται πλέον αυτό το ζήτημα. Και τέλος Πρόεδρε. Για το Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ έχω περάσει τόσο καιρό, βλέπω ότι κοιτάω τις εφημερίδες στο Ηνωμένο Βασίλειο που λένε όλη την ώρα αν θα πρέπει να μπούμε, αν πρέπει να είμαστε μέσα στην Ένωση, αν θα είμαστε έξω από την Ένωση, πώ πρέπει να περιοριστούν οι απαιτήσει. Όμως πολλές μεγάλες εμπορικές εταιρείες έρχονται και μου λένε ότι το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι 27 διαφορετικά είδη του ροζ. Θέλουμε συνεπή νομοθεσία τέτοιου είδου που μας δίνει ισότιμο πεδίο δραστηριότητας. Είναι καλό για τις επιχειρήσεις, καλό για τις θέσεις απασχόλησης και για την Ευρώπη. Ευχαριστούμε Chris Ντέβις, η Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητρία Πολύ σαφή η παρουσίαση των θέσεών της. Εγώ προσωπικά, που είμαι και νέος, νέο μέλος της Επιτροπής, έμαθα πολλά για το πώς ε, μπορεί κανείς να περιγράψει με τρόπο σαφή, προσεκτικό και κατανοητό το πώς θα προχωρήσουμε με την έκθεση αυτή. Μερικές παρατηρήσεις από την πολιτική μου ομάδα είπε ότι θέλει να διευρυνθεί ο κατάλογος με τρόπο σαφέστατο των ουσιών. Καταρχήν δεν διαφωνεί κανείς, αλλά νομίζω ότι η Επιτροπή κάνει ε, πρόταση σαφή να μην το πράξουμε ε, με τον τρόπο που θέλει η συγγήτρια επί του παρόντος. Και είναι σημαντικό αυτό όταν έρθει η έκθεση σε λίγες εβδομάδες η συγγήτρια να έχει την επιστημονική τεκμηρίωση ε, σε λεπτομέρειες ε, περιστατωμένη για να πάρουμε την απόφαση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το προτείνει αυτό. Τώρα, το κατά πόσο το ροζ επικαλύπτεται με το ΡΙΤΣ. Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει μια συνάντηση της ομάδας εργασίας στην Παρασκευή ε, που ε, θα βγάλει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για τη μεθοδολογία. Ε, είμαι βέβαια ότι τα ξέρει και η Τζίλ αυτά και με χαρά προσβλέπω στη σαφή εξήγηση στην έκθεση της για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, ο Κάρλος Σλίτερ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εισηγήτρια. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν ξαναρχίσαμε τις ιστορίες στο δικαστήριο για το 10BD και επίσης χαίρομαι για την αντιστροφή του βάρους απόδειξης που είναι η, μόνο, η μόνη λογική επιλογή. Επίσης, ε, χαιρετίζω τις προτάσεις της ε, εισηγητριάς. Επιτρέψτε μου δύο θέματα να προσθέσω. Πρώτον, ας αφήσουμε να ορθοποδήσει το ΡΙΤΣ και να, υπάρχει, να συνυπάρχει με το ΡΟΣ. Η ΕΧΑ, ο οργανισμός, τα επόμενα 11 χρόνια θα έχει πάρα πολλή δουλειά για την εφαρμογή του ΡΙΤΣ και μετά από 11 χρόνια ας δούμε. Έστω λοιπόν και το ΡΟΣ, έστω και το ΡΙΤΣ και να ζήσουν και χρόνια πολλά και ευτυχισμένοι. Τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο ε, η πρόταση είναι σκόπιμη. Είναι πολύ επιφυλακτική. Ε, θα μπορούσε να βάλει και άλλες ουσίες. Από αυτούς τους 30 λόμπις που ήρθαν σε σένα, Κρίς, ε, ποιοι ήταν οι παραγωγή, ποιοι ήταν οι καταναλωτές οι άρρωστοι που έχουν πληγεί από τις φθαλικές ουσίες, από βαρέα μέταλλα. η φωνή τους δεν ακούγεται. Ξέρω ότι εσύ τους ακούς, αλλά Α μην ξεχνάμε ότι μπορεί να λέει μερικά πράγματα βιομηχανία, αλλά αυτοί που έχουν πληρώσει την ύφη, τα θύματα, σπάνια φτάνουν στα γραφεία μα και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μα. Και για τον ιατρικό εξοπλισμό θα πρέπει να είναι η μέθοδο του ανοιχτού πεδίου εφαρμογή εδώ και ε, όταν μιλάμε για πρόσθεση ουσιών, ε, για την ε, απαγόρευση Καλό είναι να γίνει μέσω του γιατί είναι πιο εύκολο να ε, έχουμε εξαιρέσεις και παρεκκλήσεις σε σχέση με το ριτς. Προσέξτε, δεν ξέρω αν θα πρέπει να βάλουμε εδώ κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε διατήρηση, συντήρηση του παλαιού. Όταν λέμε το νέο είναι πολύ ακριβό, δεν έχει μεγάλη αγορά, δεν παράγεται σε μεγάλες ποσότητες επαρκής, ε, τότε δεν θα είχαμε περάσει ποτέ από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως στο LED. Ή προσπάθησα να αγοράσω οθόνη πέρσι για τον υπολογιστή μου. LED δεν υπήρχε πέρσι, φέτος υπάρχει. Και δεν έχει και βρωμιούχα και είναι πολύ καλύτερο για το περιβάλλον. Και δεν έχει και μόλιβδο και, ε, δεν, ε, και είναι εύκολο να αποσυναρμολογηθεί από τον υπολογιστή, αλλά δεν μπορώ να τη βρω αυτή την οθόνη που θέλω. Και τέλος για την νανοτεχνολογία, ε, γιατί δεν το βάλατε αυτό. Μου λείπει από τη λίστα, θέλω να συμπεριληφθεί. Όταν το συζητήσαμε, το Κοινοβούλιο είπε ότι η παρούσα νομοθεσία τα ρυθμίζει όλα αυτά και περίπτωση θα δούμε με μονομένες περιπτώσεις. Ορίστε, φτάνουμε τώρα στις μεμονωμένες περιπτώσεις νομοθεσίας. Αυτά τα θέματα της νανοτεχνολογίας δεν θα τα βάλουμε στο ροζ. Αυτά. Θα κάνω τροπολογίες σχετικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι λίγο μπερδεμένος. Ιδιαίτερα μετά από την παρέμβαση του κυρίου Ντέιβις, ότι δηλαδή πρέπει να παραμείνουν δύο νομοθεσίες ε, παράλληλα λειτουργώντας το ΡΙΤΣ και το ΡΟΣ. Εγώ θα ήθελα να ακολουθούσαμε περισσότερο την ε, κατεύθυνση όπου αμέσως ζητούμε μια σύγκληση Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ πως ε, το REACH ε, θα πάρει 8-10 χρόνια για να εφαρμοστεί. Εγώ δεν το δέχομαι. Ας ασχοληθούμε με αυτό το πρόβλημα και να μην κάνουμε το ροζ επειδή το REACH προχωράει πιο αργά. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ να αφήσουμε το REACH να καθυστερεί τόσο. Κάτι τέτοιο θα ήταν απαράδεκτο. Επειδή λοιπόν εγώ δεν βλέπω να υπάρχει διαφορά για, από το αν χρησιμοποιείται ένα τοξικό στοιχείο για την ηλεκτρονική ή την ηλεκτρική βιομηχανία ή αν χρησιμοποιείται αλλού ότι μπορεί να υπάρχουν διακρίσεις, ότι υπάρχει διάκριση. Εμείς τι θα κάνουμε με κάτι τέτοιο, απλώς αυξάνουμε την σύγχυση. Και για το θέμα του αποκλεισμού της, της απαγόρευσης χρήσης αυτών των προϊόντων θα πρέπει να αναφερόμαστε στη μεθοδολογία REACH. Γιατί αυτή είναι που από πρακτικής άποψης ε, δίνει την μεθοδολογία της αξιολόγησης του κινδύνου και της διαχείρισης του κινδύνου. Άρα λοιπόν πιστεύω πως ήταν σκόπιμο να αναζητήσουμε και σε αυτή τη φάση την μέγιστη δυνατή σύγκληση των δύο κειμένων, ώστε να υπάρξει σύμπραξη μεταξύ των δύο. Γιατί αν τα κρατήσουμε χωριστά θα καταλήξουμε στο να έχουν και οι δύο καθυστέρηση. Αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Βαμπρέμπτου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ με τις φιλοφρονήσεις προς την εισηγήτρια. Μπράβο της πραγματικά για τη δουλειά της προσβλέπω στην έκθεσή της, γιατί βλέπω ότι έχει τη φιλοδοξία να βελτιώσει σημαντικά και να συμπληρώσει την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση τώρα για το REACH και το ROS, πρέπει να καταλάβουμε ότι το REACH δεν μπορεί να είναι άλοθη για να μην κάνουμε αυτά που πρέπει στο ROS και τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Πολύ ωραία τα είπε ο κύριος Ντέιβις. Δυστυχώς, πολύ συχνά βλέπουμε να καταλήγουν κάποια προϊόντα εκεί που δεν πρέπει και θα πρέπει να είναι και ασφαλή. Θα ήταν κρίμα λοιπόν να μπούμε στη φιλοσοφία ότι αφού έχουμε τώρα το ρίτσε δεν χρειάζεται να ενισχυθεί το ρόστι να το κάνουμε. Όχι, είναι λάθος αυτό. Και περιμένω λοιπόν την έκθεση και περισσότερες λεπτομέρειες όταν θα την έχουμε στα χέρια μας. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Κέγκλερ και μετά στην εισηγητριά μας Παρακαλώ να μην υπερβείτε το πεντάλεπτο ο καθένα σας στις απαντήσεις, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Να εξετάσουμε. Έχετε το λόγο, κύριε Κέγκολα. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Σας ευχαριστώ όλους για τις ε, τοποθετήσεις. Ήταν πολύ διαφωτιστικά και ενημερωτικά αυτά που ακούσαμε και τη σκέψη της ηγήτριας. Ελπίζω να μην χρειαστεί να εξαντλήσω το πεντάλεπτο. Θα ήθελα να αφαιρθώ σύντομα σε δύο θέματα. Πρώτον, το θέμα του πεδίου εφαρμογή. Γνωρίζουμε όλοι βέβαια ότι το λεγόμενο ανοιχτό πεδίο εφαρμογής ε, είναι θέμα που συζητείται, αυτό το open scope. Μπορεί να φαίνεται ελκυστικό σε ορισμένους από κάποιες απόψεις. Γιατί όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το παρόν δεν είναι πεπισμένη ότι θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο και παραμένει και εμένει στην πρότασή της για τον εξή λόγο. Όταν έχει κανείς ένα περιορισμένο πεδίο εφαρμογής όπως ισχύει τώρα, κάπου πρέπει να το περιχαρακώσουμε αυτό, να τραβήξουμε μια διαχωριστική γραμμή γύρω-γύρω. Και έχουμε την εμπειρία ότι όταν ε, παραμένουμε σε πολύ αόριστες διατυπώσεις, αυτό δεν μας βοηθάει. Θα πρέπει να καταλήγουμε σε παραδείγματα. Όταν λέμε παιχνίδια, παιχνίδια τι εννοούμε, γενικά παιχνίδια, πρέπει να το συγκεκριμενοποιούμε κάπου. Επειδή το συζητώ και με άλλους, νομίζω ότι αν βάλουμε ανοιχτό πεδίο εφαρμογής, ε, δεν θα λύσει το πρόβλημα από ένα περιορισμένο ε, πεδίο εφαρμογής, θα περάσουμε σε ένα χανές, ανοιχτό και θα μιλάμε για εξαιρέσεις, οι οποίες εξαιρέσεις από εκεί και πέρα θα πρέπει να έχουν μια διαχωριστική γραμμή. Τι θα εξαιρείτε και τι όχι και γιατί. Μπορεί να σας ε, αναφέρω έτσι ξεκρέμαστη μια ιδέα ε, ηλιακοί συλλέκτες, α πούμε. Δεν είναι πολιτικό το θέμα, παράδειγμα είναι. Αν έχουμε εξαίρεση για τους ηλιακού συλλέκτες, πολύ γρήγορα θα πρέπει να ορίσετε για τι είδου συλλέκτες και πανό ηλιακά μιλάμε. Ε, αποκλείονται όλα τα παιχνίδια, οποιοδήποτε παιχνίδι ή ρολόι ή ρολόι χειρός που ε, ε λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια. Καταλαβαίνετε αυτό το παράδειγμα λοιπόν ε, όταν ε, είναι ανοιχτό το πεδίο και βάζουμε αυτούς τους περιορισμούς. Αν δεν ορίσουμε πολύ συγκεκριμένα με παραδείγματα τις εξαιρέσεις δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και κάτι άλλο που μας ανησυχεί πολύ περισσότερο, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απλούστατα στοιχεία αρκετά στη διάθεσή μας για να ξέρουμε τι σημαίνει ανοιχτό πεδίο ως προς τον γενικότερο αντίκτυπο και ε, δεν μιλώ μόνο για περιβαλλοντικό αλλά και κοινωνικό και οικονομικό. Μας υποσχέθηκαν μελέτη αντικτύπου σε ένα κράτος μέλος ε, τις επόμενες εβδομάδες. Υποτίθεται ότι είναι στο στάδιο της προετοιμασίας. Εγώ δεν θέλω να δογματίζω, αλλά προσβλέπουμε με μεγάλο ενδιαφέρον ε, στις πληροφορίες και στα στοιχεία. Αυτά για το θέμα του ανοιχτού πεδίου, μη περιορισμένου δηλαδή. Και επανέρχομαι στη διαδικασία ΡΟΣ για τον εντοπισμό μελλοντικών ουσιών που θα πρέπει να απαγορευθούν. Και πάλι θεωρώ ότι η κατάστασή μας που αντιμετωπίζουμε δεν είναι άσπρο-μαύρο. Θα το κατανοούσα, μα έλεγε ο συνομοθέτης ότι κοιτάξτε παιδιά δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, δεν σας δίνουμε λευκή επιταχή στην επιτροπολογία, την έχουμε ζήσει αυτή τη συζήτηση πάρα πολλές φορές και ε, για τα, ε, την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα. Το καταλαβαίνω, αλλά από εκεί και πέρα για τα πρακτικά της συναπόφασης και αυτά έχουν τα όρια τους. Όταν μπαίνουμε σε πάρα πολύ μεγάλες τεχνικές λεπτομέρειες και τέτοιες αποφάσεις, πώς θα γίνεται αυτό στη συναπόφαση. Και πάλι απευθύνω μία έκκληση να βρούμε τη χρυσή τομή κάπου, να βάζει το πλαίσιο συνομοθέτης πολύ συγκεκριμένα και πολύ ε, ευσυνείδητα να θέτει τα πλαίσια και τα όρια και από εκεί και πέρα οι τεχνικές λεπτομέρειες να είναι στην επιτροπολογία. Νομίζω αυτό είναι κάτι που εξυπηρετεί το πνεύμα και των δύο διαδικασιών. Αυτά προς το παρόν και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα δίνω το λόγο στην συγκήτρια, την κυρία Εβάνς, αν θέλει, να απαντήσει Σεβόμενοι το πεντάλεπτο σας παρακαλώ πολύ. Thank I, be quite brief. I think, um, Μπορώ να είμαι πάρα πολύ σύντομη. Μεγάλη συμφωνία είχαμε για κάποια θέματα όπως είναι εξαιρέσεις, περιορισμοί, η νανοτεχνολογία κτλ. Για το πεδίο εφαρμογής εξακολουθώ να πιστεύω, παρά τα όσα μας είπε τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι χρειαζόμαστε ανοιχτή, ανοιχτό πεδίο για περισσότερη σαφήνεια. Και αν κοιτάξουμε τον κατάλογο στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχουν κάποια πράγματα πολύ προφανή που λείπουν, όπως είναι οι ε, ηλεκτρικοί ε, βραστήρες, ας πούμε, ή ε, οι ηλεκτρονικές κάμερες. Υπάρχουν ας πούμε εδώ. Τώρα, για το θέμα των κοινωνικο-οικονομικών ε, κριτηρίων, στα οποία αναφέρθηκε ο Κάρλ Σλούτερ, συμφωνώ απολύτως. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί ε, αν θα πρέπει να δοθεί όχι η εξαίρεση, η παρέκκληση. Ε, οι μόνοι όροι και περιορισμοί θα πρέπει να αφορούν τη διάρκεια της εξαίρεσης και το χρονοδιάγραμμα δηλαδή ε, μέχρι να βρεθεί εναλλακτική ε, λύση και προϊόν. Τώρα, για το REACH και το ROS, το REACH είναι νόμος ε, για τα χημικά, αλλά δεν προβλέπει τι θα γίνει με τα απόβλητα, ας πούμε για τα PVC, για κάποιες ουσίες που επιβραδύνουν ε, τις φλόγες. Είναι διαφορετικό το ροζ, λοιπόν, και έχει και γενικότερη παγκόσμια ισχύ. Δεν είναι το περιφερειακό που έχει το ρίτς. Καλό είναι να διατηρεί την ανεξαρτησία του και την ύπαρξή του παράλληλα με το ρίτς και το ροζ. Θα κάνω προτάσεις και σκιώδεις ηγητές ε, προηγουμένως είπαν ότι λειτουργεί σωστά και είναι κάτι που μας χρειάζεται. Ας το αφήσουμε σε λειτουργία για να δούμε τι νέοι περιορισμοί θα χρειαστούν και να φτάσουμε πιο κοντά στους στόχους για τους οποίους ε, σχεδιάστηκε στην αρχή η οδηγία. Ευχαριστώ πολύ. Madame Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σίτρια, για την, έκθεση, την παρουσίαση αυτή. Λοιπόν, θυμίζω, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 14 Ιανουαρίου 2010 στις 6 το απόγευμα. 15-17 Μαρτίου θα συζητηθεί στην Επιτροπή, 6-7 Απριλίου ψηφοφορία στην Επιτροπή και ψηφοφορία στην Ολομέλεια το Μάιο. Σας ευχαριστώ και συνεχίζουμε με το επόμενο θέμα που αφορά τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς. Και θα δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας. Βλέπω ότι σας συναρπάζει το θέμα αυτό. Το λόγο ε- έχει η εισηγήτρια η κυρία Ντεμπρούν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τα εξηγήσω όλα αυτά ε, παρόλες τις μετακινήσεις που έχουμε εδώ πίσω ε, και το θόρυβο. Πρέπει να σας πω πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει κάποια συνεργασία ήδη για την έκθεση αυτή και είμαι πολύ ευγνώμων προς όλους εκείνους που συνεργάστηκαν μαζί μου μέχρι σήμερα. Θα εξηγήσω δύο λόγια το ιστορικό και το υπόβραθο. Υπάρχει εναρμόνιση. Thank you very much. Σας ευχαριστώ εναρμόνιση των κανόνων λοιπόν για τις λεγόμενες μη εμπορικές μετακινήσεις ζώων συντροφιάς στο EC 998 ε, του 2003. Είναι για γάτες, σκύλους, ε, παπαγάλους, όλα τα ζώα συντροφιάς που έχουν και διαβατήριο ε, και αποδεικνύει ότι έχουν κάνει αντιλησικό ορό. Επίση, και ένα μεταβατικό καθεστώς που επιτρέπει σε διάφορα κράτη-μέλη να έχουν πιο αυστηρέ ρυθμίσει ανάλογα με την νόσο. Η μεταβατική ε, διάταξη για τη Λύσα ε, κανονικά λήγει τον Οκτώβριο του 2008 έλεγε, και παρατάθηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2010 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα προτείνει να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2011 για μετακινήσεις ζών συντροφιάς και εντός της Ένωσης και από τρίτες χώρες. Και προτείνεται αυτή η μεταβατική ρύθμιση να διαρκέσει μέχρι, επαναλαμβάνω, τις 31 Δεκεμβρίου του 2011. Μετά την ημερομηνία αυτή, ε, η ημερομηνία αυτή συμπίπτει καλύτερα με την περίοδο που θα τερματιστεί και η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τον εμβολιασμό ε, με αντιλησικό ρο σε διάφορα κράτη-μέλη. Ανάλογα λοιπόν με την κατάσταση έχει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρει μέτρα για άλλες ε, νόσους, για χινοκοκίαση και για κρότονες, τσιμπούρια δηλαδή. Και υπάρχουν και ε, άλλες προτάσεις. Το σύστημα ταυτοποίησης στο άρθρο 1.1 και στο παράρτημα 1.8 όπου γίνονται προτάσεις για τον αντιλησικό εμβολιασμό και 1, 2 και 1 β το παράρτημα και η διαδικασία επιτροπολογίας αφορά ένα νέο θέμα Β2 και άρθρο 5, παράρτημα 1α, άρθρο 1.8 της πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα επανέλθω σε αυτό. Συνιστώ λοιπόν να εγκρίνουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν προτίθεμαι να κάνω τροπολογίες πέρα από τρεις τεχνικές αλλαγές που έχω στην έκθεσή μου, που είναι τυπογραφικά βασικά ε, παραγράμματα στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν δείτε τις τρεις τροπολογίες, δύο αφορούν και μόνο στη λέξη υγεία. Υγειονομικά μέτρα, ε, το ίδιο και στο 2 τα προληπτικά υγειονομικά μέτρα που αναφέρονται στο στοιχείο Β μπορούν να καθοριστούν και η τρίτη τροπολογία αφορά τα ζώα που μπαίνουν σε καραντίνα και έχουν αφαιθεί κάποια, ε, κάποιες λέξεις που λέει εκτός εάν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 6 μετά την είσοδό τους στην κοινότητα. Η πρόταση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σαφώς βασισμένη στο γεγονός ότι είναι υπέρ της αρχής προφύλαξης, παίρνουν τα μέτρα τους, καλύτερη πρόληψη επιπλέον και υγειονομικά μέτρα που έχουν να κάνουν με την ενιαία αγορά και την ελεύθερη διακίνηση και κυκλοφορία των ζώων συντροφιάς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει υπόψη και τις διάφορες ε, νομοδοτήσεις της ΕΦΣΑ και καλά κάνει και ζητάει παράταση μέχρι να τελειώσει και η χρηματοδότηση των αντιλυσικών εμβολιασμών για να μπορέσει προοδευτικά να προσαρμοστεί το σύστημα στη νέα κατάσταση. Με δύο λόγια λοιπόν προτείνω να εγκρίνουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και, ε, χαρά να απαντήσω σε ερωτήσεις σας και να ακούσω τα σχόλιά σας και από τους και ηγητές. Α, και έχω μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά, όπως σας είπα προηγουμένως, το παράρτημα 1α και το άρθρο 1.8 της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής ετέθη το ζήτημα άτυπα από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου για το πώς θα ε, αναδιατυπωθεί το παράρτημα 1 ε, με βάση το άρθρο 21.2 κτλ. Είναι ένα ζήτημα νομικό για το πώς μπορεί να αναδιατυπωθεί το κείμενο ε, ρυθμιστική διαδικασία με έλεγχο και όχι ρυθμιστική διαδικασία, κανονιστική διαδικασία σκέτο. Δεν ξέρω, θέλω να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι πιστεύει για αυτά που λέει η νομική υπηρεσία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Ντεμπρόν. Προτείνω να δώσουμε το λόγο τώρα στην κυρία Κλένης Βίλμοτ και μετά στην κυρία Κατρίν Σούγη και στο τέλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, κυρία Βίλμοτ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, διότι δεν φαίνεται να είναι επίμαχο ζήτημα. Ο κανονισμός αυτός απλά καθορίζει τους κανόνες ε, κατά τη μετακίνηση ζώων συντροφιάς ε, στα κράτη-μέλη, κυρίως ε, για την προστασία κατά της λύσας. Αναφέρθηκε η συμπεριλαμβάνει την 18, ε, παράτα... Ε, παράταση ε, για κάποια κράτη-μέλη των μεταπατικών κανόνων, η οποία θα μας βοηθήσει να υποφεληθούμε από την παρούσα εκστρατεία εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορώ λοιπόν να καταλάβω γιατί, είναι, γιατί να είναι επίμαχο το θέμα. Ξέρω ότι στις συναντήσεις των σχεδόν εισηγητών δεν υπήρχε καμία διαφωνία. Συμφωνώ με τις ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις τροπολογίες ε, της εισηγήτριας. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Σούλια. Εγώ ως και όδηση εισηγήτρια εγκρίνω την πρόταση της κυρίας Ντεμπρά. Δεν χρειάζεται να τροποποιηθεί αυτό το κείμενο πέρα από τις προτάσεις που έχουν γίνει και ευχαριστώ ιδιαίτερως την κυρία Ντεμπρά που απάντησε με υπομονή σε όλες μου τις ερωτήσεις. Υποστηρίζω λοιπόν την έκθεση της κυρίας Ντεμπρά. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκολσον ζήτησε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ μπορώ να είμαι πολύ σύντομο και να υποστηρίξω την έκθεση της εισηγήτριας. Την ευχαριστώ. Έκανα εξαιρετική δουλειά. Να πω μόνο ότι στα μήκη και στα μάκρη της Ευρώπης ε, πολλοί πιστεύουν ότι τα ζωάκια τους είναι τα πιο σημαντικά στον κόσμο και θεωρούν ότι είναι η προτεραιότητά τους. Και είμαι ευτυχής που η Κομισιόν επεκτείνει αυτή την νομοθεσία και επιτρέπει σε αυτές τις χώρες να έχουν την επιπλέον προστασία που θέλουν και ξέρω πως δεν θα ισχύσει για κάποιο χρονικό διάστημα και αλλά το μόνο ερώτημα που θέλω να ρωτήσω είναι θα Είναι καλό να εφαρμόζονται αυτοί οι πιο αυστηροί κανόνες για τα ζώα για τα οποία πάνε και έρχονται σε διάφορες χώρες. Και κυρίως σε αυτή την φάση που βρισκόμαστε στη διαδικασία προστασίας εμών των ιδίων, Θα πρέπει να τον αγνωρίσουμε το ειδικό αυτό καθεστώς και δέχομαι την πρόοδο που έχει συμβεί όσον αφορά την εκρίζωση του προβλήματος σε άλλα μέρη σε άλλα κράτη-μέλη και ελπίζω ότι μέχρι το 2011 θα έχουμε επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα της εκρίζωσης. Ωστόσο μέχρι τότε είναι σημαντικό να δεθεί αυτή η παράταση. Η εναρμόνιση είναι επιθυμητή σε αυτού του τομεί, όχι μόνο σε αυτού του τομέα, αλλά και σε άλλου τομεί. Ιδιαίτερα στου τομεί που αφορούν την υγεία των ζώων και των ανθρώπων, δεν πρέπει να κάνουμε συμβιβασμού. Εγώ δεν θέλω να υποβάλω τροπολογίε, όπω είπαμε. Και οι σκιώδει συζητητέ το, είπαν, το είπε ότι δεν υπήρχε συνένεση. Όμως, Κάναμε όλη αυτή τη δουλειά για να το παρατείνουμε μόνο για 18 μήνες. Νομίζω ότι ήταν πολλή δουλειά. Μήπως θα έπρεπε ακόμα 18 μήνες να το κρακάνουμε. Και αν τελικά όλες οι υπόλοιπες επικράτες έχουν ε, τελείως εκριζώσει τη λύση, να επανέλθουμε και βέβαια να ξανακάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Μήπως μπορεί να αναφερθεί σε αυτό το σημείο η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σνέλχαρτ. Ναι, ευχαριστώ μάλιστα. Κυρίες και κύριοι. Αυτό που προτείνει η συγγήτρια είναι καλό πιστεύω. Παρ' όλα αυτά, με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγώ έχω μερικά προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια κάναμε πολλές πρόοδους ε, στη Λίσσα αν σκεφτούμε τι γινόταν πριν από 10 χρόνια, είναι πραγματικά αλλαγή στην Έχει σχεδόν εκκριζωθεί η λύσα. Όταν κυκλοφορούν ε, και ταξιδεύουν ε, ζώα, ε, σκυλιά, γάτες. Βεβαίως θα πρέπει να ελέγχονται οι ρυθμίσεις και να εφαρμόζονται οι διατάξεις στα σύνορα. Καλό και απαραίτητο και μετά το 2011. Και τα χαρτιά και τα στοιχεία των ζώων με πολύ συγκεκριμένους κανόνες που τους έχουμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά και στην πράξη έχω ζήσει ότι ακριβώς οι χώρες αυτές, και μιλάω εδώ για τη Μεγάλη Βρετανία, που έχουν αυτή την εξαίρεση, βάζουν και επιπλέον διατάξεις και μπορούν να τις ε, αποφασίζουν. Και είναι αρκετά σκληρά τα μέτρα πολλές φορές. Αρκεί να έχει κάνει ένα λάθος ε, κτηνίατρος ε, στο έντυπο, κλείνουν σε να το ζώο έξι εβδομάδες και δεν ξέρει ο δεκτήτης τι να κάνει. Δηλαδή πώς να το ρυθμίσει, επειδή υπάρχει ένα λάθος στο έντυπο. Και μετά από έξι εβδομάδες το βρίσκει και μισό τρελό το ζώο του. Ρωτώ λοιπόν, γιατί να υπάρχει αυτή η παράταση, καλή συνοριακή έλεγχη και κανένας δεν τους αμφισβητεί, αλλά εδώ μιλάμε και ψηφίζουμε ότι κάποια κράτη πρέπει να έχουν πιο αυστηρές ρυθμίσεις. Ακούω όμως τι γίνεται με τους πολίτες και κάποιο κόσμο που ταξιδεύει με τα ζώα συντροφιά ότι τους ταλαιπωρούν πάρα πολύ και είναι υπερβολικά σχολαστική έλεγχη στα σύνορα. Μα γιατί δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα να δοθεί αυτή η παράταση. Εντάξει, θα το αποφασίσουμε, αλλά μετά τέρμα δεν θα μπορούν πλέον τα μεμονωμένα κράτη να αποφασίζουν. Την έχουμε νικήσει τη λύσα σχεδόν ε, παντού στην Ευρώπη. Είμαστε μια αγορά, δεν θα πρέπει να ζητάνε εξαιρέσεις διάφορες χώρες γιατί θέλουν έτσι με φυρμάνια να επιβάλλουν πράγματα δικτατορικά. Ο κύριος Τρεμόπουλος παρακαλώ και μετά η Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, βεβαίως αυτό το σχέδιο ε, μιλά για τους υγειονομικούς όρους ε, υπάρχει όμως μια ανάγκη να αναφερθούμε στο τι ακριβώς είναι κατοικίδιο. ακούσαμε εδώ ε, ότι περιλαμβάνει ο ορισμός και γάτες και σκύλους και παπαγάλους. Ε, μέσα στην αιτολογική έκθεση αναφέρονται οι και βλέπω ότι περιλαμβάνονται και άλλα είδη άγρια ζωής τα οποία κάποια από αυτά είτε προστατεύονται είτε πια έχουν τόση διάδοση και πάνε να γίνουν και ενδυμικά είδη σε κάποιες περιοχές ανατρέποντας ε, την υπάρχουσα ισορροπία. Από την άλλη έχουμε συνείδηση ότι περίπου το 1 τρίτο των ηχθιαλιευμάτων γίνονται τροφή για τα κατοικίδια ζώα. Υπάρχει ένα τρίτο σημείο ότι υπάρχει μια επιφύλαξη από πάρα πολλούς για τους στόχους των μετακινήσεων τουλάχιστον στην Ελλάδα έχει υπάρξει μια δημόσια αντιπαράθεση πάνω σε αυτό το θέμα και τα διατυπώνω σε αυτή τη φάση ως ε, τρία σημεία ερωτήματα με αφορμή το ε, θέμα που συζητάμε και θα ήθελα απαντήσεις. Ε, Ευχαριστώ. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Λαντομάντα. Grazie signora Presidente, grazie alla Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για την, την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε και για τα λόγια εκτίμησης προς την πρόταση της Κομισιόν. Όλες οι παρεμβάσεις υποστήριξαν την πρόταση της Κομισιόν που βασίζεται κυρίως σε ένα στοιχείο που είναι πολύ εθερετικό, δηλαδή μεγάλη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την λύσα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί όπου τα προγράμματα εκρίζωσης έχουν χρηματοδοτηθεί από την Κομισιόν και έχουν φτάσει, εκεί επετεύθηκαν πολύ, πολύ σημαντικά ε, αποτελέσματα πολύ γρήγορα που επέτρεψαν την εκρίζωση ή τουλάχιστον ε, την ε, θέση υπό στενό έλεγχο την λύσα των άγριων ζώων με θετικές συνέπειες τόσο για τα κατοικίδια όσο και για τον άνθρωπο. Ε, αυτό είναι ένα στοιχείο που θέλω να υπογραμμίσω γιατί ε, πραγματικά θα ήθελα όλες οι κοινωτικές πολιτικές να ήταν τόσο <laughs> αποτελεσματικές και τόσο επιτυχής όπως αυτή σε σχέση με τη Λύσα. Η πρόταση της Κομισιόν έχει στόχο να εναρμονίσει πλήρως το καθεστώς μετακίνησης ζώων κατοικίδιων ζώων για μη εμπορικού σκοπού. Από αυτή την άποψη θα πρέπει να είμαι ειλικρινή ότι δεν καταλαβαίνω πολύ καλά τα όσα είπε ο κύριο Σουνέλχαρτ που είπε ότι το καθεστώ που ισχύει για ορισμένα κράτη-μέλη ισχύει θα πρέπει να, να σταματήσει. Αυτό είναι η πρόταση τη Κομισιόν. Αν και η πρόταση τη Κομισιόν παρατείνει για κάποιο χρόνο το υφιστάμενο καθεστώ. Λαμβάνοντα υπόψη την ανάγκη περαιτέρω βελτίωση της κατάστασης τη λύσα σε ορισμένα κράτη-μέλη. Την ανάγκη που έχουν κάποια κράτη-μέλη επίσης που αυτή τη στιγμή χαίρουν ενό μεταβατικού καθεστώτος για να προσαρμοστούν στο νέο καθεστώς και να τεθεί πλήρως σε εφαρμογή το σύστημα, το ηλεκτρονικό μάλλον σύστημα αναγνώρισης των σκύλων και γάτων που προβλέπεται να αρχίσει να ισχύει πλήρως τον Ιούλιο του 2011. Αυτά είναι τα αίτια που οδήγησαν την Επιτροπή να παρατείνει για ένα σύντομο χρονικό διάστημα το μεταβατικό αυτό καθεστώς, αλλά με τη διευκρίνηση πως αυτό το μεταβατικό καθεστώς θα πρέπει να φτάσει και στο πέραστο. Όσον αφορά τα άλλα επιχειρήματα που έθιξε ο κύριος Τρεμόπουλος, πιστεύω πως σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν το πεδίο εφαρμογής αυτής της πρότασης της Κομισιόν που αφορά αποκλειστικά την μετακίνηση για μη εμπορικούς σκοπούς κατοικίδιων ζώων. Η Κομισιόν έχει εργαστεί ιδιαίτερα σε σχέση με τις ε, υδατοκαλλιέργειες και με την πολιτική της ε, υγείας των ζώων για τα ζώα τα υδρόβια. Έχουμε μια νέα οδηγία τη 2006-88 σε σχέση με τα ζώα της και την υδατοκαλλιέργεια. Έχουμε εφαρμόσει μια σειρά μέτρων σε σχέση με αυτή την οδηγία ακριβώς μέσα στο 2008 και το 2009 και σε σχέση με τη χρήση των ηχθιάλευρων έχουν γίνει πολλές αλλαγές κατά τη διάρκεια της πρόσφατης, ε, του πρόσφατου κανονισμού για τα υποπροϊόντα που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και που θα δημοσιευθεί εντός ολίγου στην επίσημη εφημερίδα για τον οποίο ήταν εισηγητής ο κύριος Νέλχαρντ κατά τη διάρκεια της περασμένης θητείας. Όσον αφορά το θέμα τώρα της εισηγήτριας σε σχέση με τις πτυχές της επιτροπολογίας θα ήθελα να δώσω το λόγο, αν η πρόεδρος μου το επιτρέπει, στη συνάδελφο Άννα Μαρκούλη της νομικής υπηρεσίας που θέλει να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα της εισηγήτριας. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Ευχαριστώ. As, you 1A. Όπως βλέπετε το παράρτημα 1α της πρότασης ε, περιλαμβάνει σαφώς τεχνικούς κανόνες, πιο συγκεκριμένα οι τεχνικοί προσδερισμοί για τους μεταφορείς. Η Κομισιόν θέλει να επιστήσει την προσοχή σας στο γεγονός ότι αν κάποιος δει τα άρθρα 4α και 13 όπου γίνεται η αναφορά στις απαιτήσει αυτού του παραρτήματος θα, δούμε, θα δει μάλλον ότι αν οι απαιτήσει του παραρτήματος 1α δεν τηρηθούν τότε ο ιδιοκτήτης του κατοικιδίου εξακολουθεί να μπορεί, να, να μάλλον να μάλλον εξακολουθεί να οφείλει να δώσει ε, διαβεβαιώσεις για την ανάγνωση αυτού του στοιχείου μεταφοράς. Δηλαδή δεν μιλάμε για αυστηρά δεσμευτικούς κανόνες στο παράρτημα 1α. Θέλουμε επίσης να διευκρινίσουμε πως αυτή ήταν μια ξεκάθαρη βούληση της Κομισιόν να προβλέψει έτσι ώστε η σύνταξη αυτών των κανόνων να γίνεται μέσω της ε, φυσιολογικής ρυθμιστικής διαδικασία. Θα θέλαμε επίσης να επιστήσουμε την προσοχή σας στο άλλο παράρτημα που εισάγεται μέσω αυτής της πρότασης, σύμφωνα με το οποίο βλέπουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για τον εμβολιασμό κατά της λύσας, αυτό το παράρτημα θεωρήθηκε ότι έπρεπε να περάσει από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και γι' αυτό με βάση μάλλον αυτήν την λογική η Κομισιόν αποφάσισε αυτά τα καθαρά, αυτά τα καθαρό, καθαρά τεχνικό παράρτημα το 1α να παραμείνει στην απλή ε, ρυθμιστική διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για πολύ λίγα λεπτά η Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πολύ λίγα λεπτά μόνο. Αν μου επιτρέπετε, ευχαριστώ όλους τους κοιόδης ηγητές και τα υπόλοιπα μέλη που μίλησαν για τα καλά τους λόγια. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απάντησή της στην ερώτησή μου. Πιστεύω και εγώ ότι το πεδίο της δικής μου έκθεσης δεν μπορεί να καλύψει όλα τα θέματα ε, που ε, ε, ρωτήθηκαν γιατί μιλούμε για τη μη εμπορική μεταφορά. Τώρα, για το χρονοδιάγραμμα που έθεσε και ο κύριος Νίκολσον και ο κύριος Σνέλχαρτ, φαίνεται από τις εκθέσεις της ΕΦΣΑ ότι υπάρχει ένας επιπολασμός της λύσας σε κάποια κράτη-μέλη και βάσει αυτών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει προγράμματα με υποστήριξη κοινοτική και είναι σωστό αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταβατικό αυτό μέτρο να παραταθεί μέχρι να έχουν φτάσει στο στόχο τους και τα προγράμματα αυτά. Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις που μπορεί να κάνατε, αλλιώς με χαρά να συζητήσουμε όποτε θέλετε για να σας δώσω οποιαδήποτε διευκρίνηση ενημερώσει. Ευχαριστώ κυρία εισηγητρία για την εργασία σας. Θυμίζω τις προθεσμίες. Κατάθεση τροπολογιών 9 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Ψηφίζουμε την 1η Δεκεμβρίου εδώ στην Επιτροπή. Η Ήτρε, συγγνώμη, διορθώνει η Πρόεδρος γιατί μιλάει για άλλο θέμα. Λοιπόν, 11 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, 12 το μεσημέρι και 1 Δεκεμβρίου ψηφίζουμε. Ε, αυτές οι ημερομηνίες. 11, 11 και 1η Συνεχίζουμε. Επενδυτικά σχέδια σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ένα τέταρτο θα παρακαλούσα να ασχοληθούμε με το κείμενο αυτό, γιατί μετά δείτε τι έχουμε. Διάθεση στην αγορά και χρήση των βιοκτώνων που είναι ένα θέμα πιο μακροσκελές και θα δώσω αμέσω το λόγο στον κύριο Πηδίγιο. Αν μπορείτε ένα πεντάλεπτο θα ήταν θαυμάσιο. Farò più breve possibile, signora Presidente, onorevoli colleghi. Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν, αγαπητοί Πρόεδρε και συνάδελφοι. Το νέο σενάριο ενεργειακής πολιτικής και οι πολιτική στόχοι για ε, το ενεργειακό μίξε θα οθήσουν τους φορείς σε διάφορες νέες επενδύσεις στι υποδομέ για την ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωση. Η πρόταση κανονισμού για την κοινοποίηση για την ευρωπαϊκή την Ευρωκομισιόν ε, για αυτά τα προϊόντα, για μάλλον αυτά τα προγράμματα που είναι ο 732 97 θα επιτρέψει την Επιτροπή να έχει στοιχεία και πληροφορίες για τα προγράμματα επενδύσεων των κρατών μελών που αφορούν, αφορούν την παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου, παραγωγή βιοκαυσίμων και εγκαταστάσεις αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα. Οι διευκρινήσεις όσον αφορά αυτές τις πληροφορίες θα επιτρέψουν στην Κομισιό να παρακολουθεί στην κατάσταση της ενέργειας και να έχει ένα πλαίσιο όσο γίνεται, πιο, ε, όσο γίνεται πληρέστερο όσον αφορά τις ε, παραγωγικές δυνατότητες των διαφόρων εγκαταστάσεων και να επιτρέψει έτσι μια σύγκριση και μια αξιολόγηση για την ε, προσφορά και τη ζήτηση στην ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κανονισμός αποτελείται από 13 άρθρα και ένα τεχνικό παράρτημα όπου αναφέρονται οι διάφοροι τύποι επενδύσεων που πρέπει να κοινοποιούνται. Με βάση τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 6 του κανονισμού, τα στοιχεία που θα πρέπει να μεταβιβάζονται θα δίνονται ομαδοποιημένα και όχι εμπορικά ευαίσθητα Εκεί η Κομισιόν αναλαμβάνει να τα δημοσιεύει. Στο άρθρο 2 δίνονται μια ολόκληρη σειρά από ορισμούς ε, για να είναι έτσι ομοιογενής η ερμηνεία όσον αφορά τις πληροφορίες που θα πρέπει να διαβιβάζονται. Η κοινοποίηση αφορά, και αυτό θέλω να το τονίσω, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 5, δεν αφορά μόνο τα επενδυτικά προγράμματα, αλλά και ενδεχόμενες, ενδεχόμενες ε, Καταργήσει διαφόρων εγκαταστάσεων. Αυτό εδώ έχει περισσότερο διοικητικό χαρακτήρα, αλλά θέλησα να υποβάλω τροπολογία στο άρθρο 5 που προβλέπει την διαβίβαση στοιχείων για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο για αυτά τα ενεργειακά προγράμματα, ώστε να είμαστε βέβαιοι ώστε, ε, ότι αυτά τα προγράμματα δεν βλάπτουν το περιβάλλον. Πάντα στο άρθρο 5, όσον αφορά τη διαδικασία κοινοποίηση για την κατάργηση χρήση υφιστάμενων ε, εγκαταστάσεων, θεωρώ πω είναι απαραίτητο η κοινοποίηση να συνοδεύεται πέρα από την κοινοποίηση τη ε, προτινόμενη κατάργηση, προβλέπεται από την προερώταση και την ενημέρωση για το σχέδιο της σταδιακής κατάργησης λειτουργίας της εγκατάστασης. Επίσης, έχω κάνει και μια τροπολογία στη πέμπτη παράγραφο σημείο 2 του πρώτου άρθρου του κανονισμού που σχετίζεται με την αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα. Η πρόταση κανονισμού προβλέπει την κοινοποίηση των ε, χώρων όπου μπορούν να αποθηκευθούν ε, πάνω από 100, ε, πάνω από 100 εκατομμύρια τόνοι. Εκεί νομίζω θα πρέπει να παρακολουθούμε τι γίνεται για να βλέπουμε ποιε είναι οι εξελίξει σε σχέση με τις δυνατότητε τη νέες τεχνολογίες αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα, ώστε να μην οδηγούμαστε σε αύξηση κόστους του για τους φορείς του για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να παρατηρήσω ότι η κοινοτική νομοθεσία που ισχύει αυτή τη στιγμή επιβάλλει ήδη υποχρεώσει ενημέρωση και κοινοποίηση όσον αφορά τι επενδύσει στι ενεργειακές υποδομέ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εγγυηθούμε ότι η έγκριση τέτοιων πληροφοριών θα αποτελεί αντικείμενο ενός καλύτερου συντονισμού έτσι ώστε να αποφευθούν επικαλύψεις όσον αφορά την υποχρέωση ενημέρωσης. Με χαρά δέχομαι και ενσωματώνω στην εκθεσή μου ενδεχόμενες προτάσεις από πλευρά των συναδέλφων. Πρόεδρε, τα είπα και γρήγορα τα συνοψίσατε, έχετε αυτή την ιδιότητα. Ο κύριος Βάλτσο έχει το λόγο. Λόγω του περιορισμένου χρόνου δεν θα μπω στα θεμελιώδη ζητήματα, θα αναφερθώ μόνο στο σχέδιο έκθεσης και τις τροπολογίες. Υπάρχουν, ε, προτείνονται κάποιες αιτιολογικές σκέψεις, από τις οποίες προκύπτει ότι η συνέπειες για το περιβάλλον θα πρέπει να αποτελέσουν το επίκεντρό μας. Ένα παράδειγμα είναι η επιθυμία ενημέρωσης σχετικά με την παρούσα υποδομή. Γιατί όμως δεν απαιτούμε περισσότερες πληροφορίες. Θα πρέπει οι πληροφορίες να φτάνουν μέχρι τους διάφορους φορείς. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν επενδύουν, όταν δημιουργείται υποδομή, για τις μεταφορές για παράδειγμα, θα πρέπει αυτό να γίνεται γνωστό. Αυτές οι πληροφορίες θα ήταν αρκετές. Ταυτόχρονα αναφέρεται ότι κατά τον παροπλισμό θα πρέπει να γίνεται περιβαλλοντική μελέτη των επιπτώσεων. Πέρα από αυτό, ζητείτε μελέτη σχετικά με τα μέτρα για τον περιβαλλοντικό τομέα. Αν κοιτάξει κανείς τους αρχικούς στόχους, θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. παράλληλα πραγματοποιούνται όλα αυτά, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο δυναμικό που υπάρχει. Και επίσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο 5, όπου αναφέρονται οι προγραμματισμένες επενδύσεις και όπου αναφέρεται η αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Θα ήθελα εδώ να ξέρω για πόσες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μιλάμε και μπορούμε να έχουμε τις ίδιες απαιτήσει στην περίπτωση πυρηνικής εγκατάστασης. Να γίνεται ενημέρωση δηλαδή σχετικά με τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων, ώστε να έχουμε επισκόπηση των προγραμματισμένων μέτρων. Παρακαλώ ε, να μιλάτε δύο λεπτά ο καθένας, αν είναι δυνατό. Κύριε Πρόντι. Θα είμαι συντομότατος, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ τον συνάδελφο Πυρίλο και συμφωνώ με τις τροπολογίες του. Μου θέλω μόνο να μιλήσω σε σχέση με την προηγούμενη παρέμβαση ότι η Κομισιόν θα πρέπει να μας πει τι θα γίνει με αυτή την κοινοποίηση. Τι θα τα κάνει αυτά τα στοιχεία δηλαδή. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πρωτοβουλίες που πρέπει να γίνουν για να βελτιστοποιηθεί η χρήση των ενεργειακών πόρων ώστε να μεγιστοποιηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να αυξηθεί η παραπληρωματικότητα των διάφορων ειδών ενέργειας. Να σας δώσω το παράδειγμα ότι τις πιθανότητες να χρησιμοποιηθεί η ολική ενέργεια μαζί με την ε, υδραυλική ενέργεια για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε το, στο, συνολικά την μεγαλύτερη δυνατή ε, εκμετάλλευση, ωφέλεια μάλλον από την ανανεώσιμη ενέργεια. Και με εγγύηση μιας συνέχειας για την παροχή ενέργειας. Όλο το θέμα λοιπόν της βελτιστοποίησης, το, της χρήσης των ενεργειακών πόρων, για παράδειγμα συν, ε, ε, συνδυασμένη ε, χρήση διαφόρων ενεργειών, θα πρέπει να προωθηθεί. Γι' αυτό και θα πρέπει η Κομισιόν να μας εξηγήσει τι θα τις κάνει όλες αυτές τις πληροφορίες. Και ποια μέτρα θα μπορέσει να λάβει ώστε να βελτιώσει την γενικότερη συμβατότητα. Ώστε το ηλεκτρικό δίκτυο να να ανταποκρίνεται στα αιτήματα και το δίκτυο φυσικού αερίου να μπορέσει να προσαρμοστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριος Εκούτου. Ευχαριστώ κύριε μου. Και συνεχίζω στα αγγλικά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον εισηγητή για την γνωμοδότησή του. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ακριβώς αναφερόμενος στο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Τα επόμενα χρόνια οι υποδομές ενεργειακές και επενδύσεις είναι κρίσιμες για να περάσουμε στους ανασιώσιμους στόχους, ε, όχι μόνο για το 2020, αλλά και πιο μακροπρόθεσμα, όταν θα περάσουμε στη μεγάλη αλλαγή και μετάβαση προς τις ανανεώσιμες. Χρειαζόμαστε κρίσιμες λοιπόν επενδύσεις και ιδιαίτερα στα δίκτυα, στο grid, ε, το ηλεκτρικό, ε, στις διασυνδέσεις κτλ. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να διατηρήσουμε την υποστήριξη που έχει ο κόσμος ε, προς αυτές τις επενδύσεις και να γίνουν χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον. Επίσης, πολύ μεγάλη σημασία έχει και το θέμα των επιλογών. Αν θα πρέπει να αντικαταστήσουμε τις υποδομές και να επενδύσουμε σε νέες ή να εξυγχρονίσουμε τις παλιές. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει και εμάς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι και πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Δεν έχω να προσθέσω και πολλά. Ένα μόνο στοιχείο επιπλέον για την ποιότητα και τη δημοσιότητα των στοιχείων του άρθρου 6 και θα πρέπει να ξέρουμε πόση διαφάνεια θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα στοιχεία. Τώρα εδώ λέει ότι δύναται να τα δημοσιεύει. May publish. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να είναι δύναται, αλλά οφείλει. Όχι may, αλλά should. Για η Ευρώπη ολόκληρη να έχει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εισηγητής μας, θέλετε το λόγο κύριε εισηγητά να απαντήσετε σε αυτές τις παρατηρήσεις proprio in qualche attimo e al primo Μια στιγμή θα πάρω μόνο. Το, το πρώτο μιλητή ζητώ συγγνώμη γιατί δεν είδα το, δεν, δεν συγκράτησα το όνομά του. Αλλά θέλω να πω ότι ότι ο κατάλογος των μέτρων που προβλέπονται για την περιβαλλοντική εξυγίανση ε, θα πρέπει να απαιτείται από τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Έχω εδώ μπροστά μου τον κανονισμό ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι προβλέπεται ε, για αυτή τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Γι' αυτό και η κάψη στην οποία αναφέρθηκε ο συνάδελφος που παρενέβη πρώτος νομίζω ότι μπορεί να ξεπεραστεί με αυτήν την πρόβλεψη εδώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο πρώτη. Ωστόσο, νομίζω πως το πρόβλημα στο οποίο αναφέρθηκε είναι πολύ πιο περίπλοκο. Η Κομισιόν θα πρέπει όντως να ασχοληθεί για να μας δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις, συμπληρώνοντας ε, αυτή τη γνωμοδότηση που, όπως όλοι γνωρίζετε, ε, πάει για την Ήτρη. Για το τελευταίο παρατήρηση για το άρθρο 6. Εγώ έχω την εντύπωση πως το άρθρο 6 είναι εξαιρετικά σαφές, διότι εδώ αναφέρεται ανάγκη δημοσίευσης των στοιχείων. Αλλά ας ε, υποθέσουμε ότι σε, μια, ένα κράτος, σε μια χώρα, υπάρχει μόνο μια επιχείρηση που κάνει μια παρέμβαση και μια τέτοια μοναδική παρέμβαση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα γιατί έτσι τα στοιχεία, αν είναι ευαίσθητα, δεν μπορούν να αποκαλυφθούν. Θα αποδοθούν σε αυτόν που κάνει την παρέμβαση, την επένδυση. Γι' αυτό λοιπόν και προσπαθήσαμε να το καλύψουμε με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ. Merci, monsieur le Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Σιγητά για αυτή τη δουλειά, για αυτή την εργασία σας. Να θυμίσω το χρονοδιάγραμμα. 9 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι για τις τροπολογίες. Ψηφίζουμε εδώ την 1η Δεκεμβρίου και στην Ήτρε 27 ε, Ιανουαρίου και στην Ολομέρεια το Φλεβάρι του 2010. Καλώς. Θα περάσουμε λοιπόν τώρα αν θέλετε, στο θέμα των βιοκτώνων, θα δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτώνων. Η εισηγήτρια είναι η κυρία Κλάς, έτσι. Η κυρία Κρίστα Κλάς, παρακαλώ. Pour votre Για μας παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μου είπαν ότι η Κομισιόν θα έχει πρώτα τη δυνατότητα να παρουσιάσει την έκθεση, την πρόταση τη Κομισιόν. σω καλύτερα να τα ακούσουμε με αυτή τη σειρά. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να μιλήσει πρώτη η Κομισιόν. Uh, Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε συντομία την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κανονισμό για τα βιοκτώνα. Περιληπτικά, η πρόταση κανονισμού στοχεύει να οικοδομήσει πάνω στα στοιχεία που λειτουργήσαν καλά κατά τα 8 χρόνια εφαρμογής ε, του παρόντος κανονισμού, τα οποία θα πρέπει να διατηρήσουμε. Η πρόταση αυτή όμως, ε, για προφανείς λόγους, θα πρέπει να αναθεωρήσει και όλα τα στοιχεία που δεν λειτουργήσαν καλά. Και θα πω σε λεπτομέρειες. στόχος της αναθεώρησης αυτής είναι διτός. Αφενός να προστατεύσουμε περαιτέρω το περιβάλλον, σημαντικό στοιχείο. Η παρούσα οδηγία ήδη έχει πετύχει υψηλό επίπεδο προστασίας ε, του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Θεωρήσαμε όμως ότι είναι απαραίτητο να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την κατάσταση και να κλείσουμε κάποια παραθυράκια που υπάρχουν ε, στην παρούσα νομοθεσία. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος βασικός στόχος. Ο δεύτερος βασικός στόχος που είναι επίσης πολύ σημαντικός, είναι να μειωθεί το παρόν υψηλό κόστος συμμόρφωσης που, που ε, αποτελεί συνέπεια της παρούσας οδηγίας, διατηρώντας όμως ε, το υψηλό επίπεδο προστασίας για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η μελέτη επιπτώσεων εξέτασε διάφορες λύσεις και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι Όλοι οι τομείς πολιτικής και όλες οι λύσει που επιλέξαμε στοχεύουν στη μείωση του κόστους για τη βιομηχανία, εκτός από μία μικρή περίπτωση που συνδέεται ε, με ε, κάποια εξαρμαζά αντικείμενα, στα οποία όμως θα, θα επανέλθω αργότερα. Στόχος λοιπόν ήταν να μειώσουμε το κόστος για τη βιομηχανία. Η πρόταση επίσης ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές από άλλα νομοθετήματα, ε, αυτό για τα παρασιτοκτόνα, το REACH και σε κάποιο βαθμό τον κανονισμό ε, ΕΜΕΑ. Να αναφερθώ στους δύο βασικούς στόχους, ε, την προστασία του περιβάλλοντος και το κόστος. Για την περιβαλλοντική προστασία είναι σημαντικό το θέμα των επεξεργασμένων προϊόντων, ε, διότι αυτή τη στιγμή μπορεί να εισάγει κανείς προϊόντα τα οποία έχουν τύχη επεξεργασίας ε, με ουσίες που απαγορεύονται στην Ευρώπη, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί αυτό. Πέρσι είχαμε περιπτώσεις καναπέδων και υποδημάτων που δημιούργησαν αλλεργίες και εγκάβματα στους καταναλωτές που, έπρεπε, που κατέληξαν ακόμα και στο νοσοκομείο. Αυτό με την παρούσα ε, πρόταση δεν θα, γίνει, δεν θα γίνεται στο μέλλον, διότι όλα τα προϊόντα που έχουν τύχει επεξεργασίας με βιοκτόνες ουσίες πρέπει να ε, έχουν ε, τη σχετική επισήμανση. Και θα πρέπει να είναι εγκεκριμένε οι βιοκτόνε ουσίε. Αυτό που συνέβη με του καναπέδε και με τα παπούτσια, με τι μπότε, ήταν ότι οι ουσίε αυτέ ήταν απογορευμένε στην Ευρώπη. Πρόκειται λοιπόν για ένα παραθυράκι το οποίο πρέπει να κλείσουμε για να έχουμε καλύτερη προστασία τη ανθρώπινη υγεία. Αυτό λοιπόν ω προ τα προϊόντα ε, τα επεξεργασμένα. Ε, Επίση έχουμε μια διάταξη για το κριτήριο αποκλεισμού, το οποίο σημαίνει ότι οι ιδιαίτερα επικίνδυνε ουσίε δεν μπορούν πια να ε, εγκριθούν, εκτός από πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, που αναφέρονται ρητά στην πρόταση. Οι πιο επικίνδυνες ουσίες όμως ε, αποκλείονται. Άλλο σημαντικό στοιχείο για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η συγκριτική αξιολόγηση που είναι πάρα πολύ σημαντική διότι βασίζεται στην αρχή της υποκατάστασης. Δηλαδή κάθε προϊόν που περιέχει ουσίες οι οποίες είναι υποψήφιες για υποκατάσταση θα πρέπει να συγκρίνονται με άλλες ουσίες ε, για να εγκριθούν. Και έτσι σκοπεύουμε να αποκλείσουμε από την, αγορά σταδιακά όλα τα προϊόντα με τις πιο επικίνδυνες ουσίες. Αυτά λοιπόν ήταν σύντομα τα θέματα που αφορούν την ε, προστασία του περιβάλλοντος. Μπορούμε βέβαια να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες ε, αν απαιτηθεί κάτι τέτοιο. Όσον αφορά την καλύτερη αποτελεσματικότητα και μείωση του κόστους για την έγκριση των προϊόντων, να σας θυμίσω σύντομα ότι ο κανονισμός ε, για τα βιοκτώνα είναι διτός. Από τη μία υπάρχει η έγκριση της ουσίας και κατόπιν η έγκριση του τελικού προϊόντος που διατίθεται στην αγορά που περιέχει την δραστική ουσία. Το ίδιο για τα παρασιτοκτόνα. Όσον αφορά λοιπόν το κόστος ε, για την ε, βιομηχανία ε, για την έγκριση των προϊόντων, η πρόταση απλοποιεί όλες τις διαδικασίες, κάτι που θα αυξήσει την νομική βεβαιότητα για τις επιχειρήσεις. Ε, εντύπωση μου κάνει ότι αυτή τη στιγμή στην παρούσα οδηγία δεν υπάρχει προθεσμία για το κράτος μέλος να εγκρίνει ένα προϊόν. Δεν υπάρχει καμία προθεσμία. Φυσικά τα κράτη-μέλη δεν περιμένουν χωρίς λόγο, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό για να υπάρχει νομική βεβαιότητα ε, να μπορεί να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις λίγο πολύ το χρονοδιάγραμμα για την τελική έγκριση ενός προϊόντος. Αυτό αφορά την ε, έγκριση των προϊόντων γενικά. Για να απλοποιήσουμε περαιτέρω το σύστημα και να μειώσουμε το κόστος, προβλέπεται κεντρική έγκριση που θα γίνεται από την ΕΚΑ, την, ε, τον οργανισμό στο Ελσίνκι. Προτείνουμε αυτό να γίνεται για τα προϊόντα χαμηλού κινδύνου καθώς και για τα προϊόντα που περιέχουν τις νέες ουσίες που θα διατίθενται στο μέλλον στην αγορά. Επίτηδες ε, περιορίσαμε περιοριστήκαμε σε δύο κατηγορίες για να δούμε αφενός σε τι βαθμό θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο για τα προϊόντα χαμηλού κινδύνου. Υπάρχουν δύο λύσεις για τις επιχειρήσεις. Μπορούν είτε να ακολουθήσουν την κανονική ε, διαδικασία μέσω των κρατών μελών, είτε να ε, χρησιμοποιήσουν τον οργανισμό ΕΚΑ. Για τις νέες ουσίες είναι σημαντικό για μας ε, να καταλήξει κανείς απευθείας στην κεντρική διαδικασία. Και σημαντικό είναι ο οργανισμός ΕΚΑ να έχει το δυναμικό για να μπορεί να ενεργήσει αποτελεσματικά στα πλαίσια του συστήματος αυτού. Επίσης, για την ε, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα έχουμε απλοποιήσει όλες τις διατάξεις που έχουν να κάνουν με την αμοιβαία αναγνώριση, ώστε ο βιομηχανικός τομέα να μην χρειάζεται να ζητήσει έγκριση σε κάθε κράτο μέλο για το τελικό προϊόν. Εάν ε, μια επιχείρηση επιλέξει να ε, ζητήσει έγκριση ενός προϊόντος σε ένα κράτος μέλος, τα άλλα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, εγκρίνουν επίσης αυτομάτως το προϊόν αυτό, εκτός αν έχουν πολύ καλούς λόγους. Η αμοιβή αναγνώριση λοιπόν υποθέτω θα λειτουργήσει καλύτερα και η διαδικασία στην πρόταση είναι πολύ πιο σαφής Επίσης, ε, Είχαμε και το θέμα των δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα, τις απαιτήσει για δεδομένα για κάποιες επιχειρήσεις. Ε, δεν χρειάζεται οι επιχειρήσεις να υποβάλουν όλα τα δεδομένα για το προϊόν και αυτό διευκρινίζεται καλύτερα στην πρόταση. Και επίσης υπάρχει διάταξη για εναρμονισμένη δομή τελών στα κράτη-μέλη. Έχουμε επίση την αρχή μείωση των τελών για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, διότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα το γεγονό ότι πολλέ επιχειρήσει είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ένα από τα στοιχεία της μελέτης επιπτώσεων ήταν ότι το παρόν κόστος υπό την παρούσα οδηγία μπορεί να βλάψει με δυσανάλογο τρόπο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις μικρές επιχειρήσεις. Και τέλος, ε, την οδηγία την κάναμε κανονισμό για να εξαλείψουμε την ανάγκη μεταβατικής περίοδου αλλά και πιο σημαντικά για να αποφύγουμε το διοικητικό φόρτο που συνδέεται με τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία. Ακόμα πιο σημαντικά όμως για να διασφαλίσουμε την ε, ε, ενιαία, την ομοιόμορφη ε, εφαρμογή. Σε μια διαδικασία όπου είναι σημαντικό να υπάρχουν σαφείς προθεσμίες και σαφείς ορισμοί. Τέλος, να πω ότι Οι τροποποίησει ε, στην ε, διαδικασία που προτείνεται στην πρόταση αυτή έχουν να κάνουν κυρίως ε, με την έγκριση των ουσιών. Η διαδικασία που ακολουθείται θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι να ολοκληρωθεί αναθεώρηση για να υπάρχει ίση μεταχείριση των παραγωγών δραστικών ουσιών η θελημένα δεν αλλάξαμε τον τρόπο που εγκρίνονται οι ουσίες. Διατηρήσαμε δηλαδή το ίδιο σύστημα που υπάρχει σήμερα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μείωση του κόστους και υψηλή, υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, όπως σας είπα νωρίτερα. Θα κλείσω εδώ, ενδεχομένως να έχω τη δυνατότητα να δώσω διευκρινήσεις, αν είναι κάτι τέτοιο απαραίτητο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έχει τώρα το λόγο, κυρία Κλάς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσίασε σε συντομία το εκτενέστατο αυτό έγγραφο και σας ευχαριστώ που έχουμε την ευκαιρία σήμερα να το συζητήσουμε αυτό χωρίς ακόμα να υπάρχει ε, έκθεση ή κανένα άλλο έγγραφο. Αυτό που με ενδιέφερε εμένα κυρίως ήταν να δω λίγο να βολιδοσκοπήσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε ε, τον κόσμο για τα βιοκτώνα. Και χαίρομαι που προχωρούμε σε βελτίωση και ε, κλείνουμε και τα ελλείμματα που είχε αφήσει η οδηγία, γιατί από το 98 και μετά έχουμε ένα κείμενο αρκετά κακογραμμένο καμιά φορά, με πολλή γραφειοκρατία και περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία έγκρισης και αδειοδότησης. Χαίρομαι που αναθεωρούμε τώρα το έγγραφο, γιατί ήταν πάρα πολλά τα σφάλματα. Τώρα την Άνοιξη αποφασίσαμε μόλις ε, παράταση των προθεσμιών μέχρι το 2014 για την αδειοδότηση, ακριβώς γιατί εδώ είχαμε μεγάλα ε, προβλήματα ε, χρονικά και μεγάλα αναμονή ε, και μποτιλιάρισμα ουσιαστικά από τις αιτήσει. Θα πρέπει να δούμε τι σημαίνουν τα βιοκτώνα για την κοινωνία. Είναι αναπόφευκτα και ε, για να διατηρήσουμε και τους όρους υγιεινής. Ε, ξεπλάγει πάρα πολύ. Παντού τα βλέπεις και αυτό βιοκτόνο είναι. Είμαστε πολύ υπέρ της υγιεινής, της προσωπικής και στο κοινοβούλιο και εδώ μέσα έχει βιοκτόνα. Ε, απανταχού παρόντα είναι και τμήμα της ζωής μας. Και πλέον στοιχείο του πολιτισμού μας ως απολυμαντικά ή ε, φυτοφάρμακα μας προστατεύουν από επικίνδυνες ε, ασθένειες και τη μετάδοσή τους. Και η κοινωνία μας απαιτεί, ακριβώς επειδή είμαστε πολύ πυκνοκατοικημένες χώρες, ιδιαίτερους όρους υγιεινής για να μην μεταδίδονται μικρόβια και αρρώστιες. Έχουμε διεθνή κινητικότητα και έτσι διαδίδονται πιο εύκολα νοσήματα ή και μικρόβια ε, αστραπία σε όλο τον κόσμο και ελπίζω να ξεπεράσουμε και το θέμα της γρήπης. Ε, η βιομηχανική παραγωγή τροφίμων και αυτή χρειάζεται συντηρητικά για να διατηρούνται τα τρόφιμα και να διατίθενται περισσότερο διάστημα. Επίσης θα πρέπει να καθαρίζονται και να πολυμένονται εργοστάσια ή ακόμα και νοσοκομεία. Ε, και θα πρέπει όλα τα πλυντήρια και καθαριστήρια να ε, καθαρίζουν και να απολυμένουν από κάθε μικρόβιο. Όλα αυτά είναι βιοκτώνα και επίσης και ως προστατευτικά ε, υλικά για το ξύλο, για ίνες, για μέσα επεξεργασίας μετάλλου, ακόμα και στους τείχους, παντού. Ε, ναι, είναι επικίνδυνα. Τι να κάνουμε, είναι δηλητήρια. Αφού σκοτώνουν ε, ε, τα παράσιτα, τα μικρόβια, ε, τους μύκητες. Γι' αυτό είναι επικίνδυνα, γιατί πρέπει να σκοτώνουν βλαβερούς οργανισμούς και θα πρέπει να είναι δραστικές ουσίες, εξού και επικίνδυνες πολλές φορές. Γι' αυτό χρειαζόμαστε καλύτερη ρύθμιση, πιο αυστηρή, να ε, ζυγίζουμε πολύ καλά το όφελος και τον κίνδυνο και δεν θα πρέπει να έχουμε πληθωριστική αλόγιστη χρήση, πάντα με ε, υπευθυνότητα. Όχι όσο περισσότερο τόσο καλύτερα, όχι, γιατί όσο περισσότερο μπορεί τελικά το φάρμακο να γίνει φαρμάκι. Ε, και χρειαζόμαστε μια στρατηγική για αηφόρο χρήση των βιοκτώνων και για εναλλακτικές ουσίες. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως δεν είναι να προστατευόμαστε από τα βιοκτώνα, αλλά να προστατευόμαστε με τη χρήση των βιοκτώνων. Όταν κάποιος έχει ψήρες, ε, κάπως θα πρέπει να τις σκοτώσει. Αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να βάλεις και τη χτένα και να ψηρίσεις ε, πριν ε, ρίξεις τη σκόνη για τις ψήρες. Στην αρχή της δεκαετίας του 80 θυμάστε ότι είχε γίνει ένα σκάνδαλο με κάποιες ουσίες προστατευτικές για το ξύλο ε, και προχωρήσαμε σε νέα νομοθεσία. Καλό είναι αυτό, χρειαζόμαστε ε, νέα προϊόντα που να σέβονται το περιβάλλον. Έχουμε νέες τεχνολογίες που λέγονται νάνοτεχνολογίες πλέον. Και θα πρέπει να είμαστε πάντα αυστηροί και επικριτικοί, γιατί όμως και τα νάνο-σωματίδια διαπερνούν και το δέρμα και το νερό θα πρέπει να υποστηρίζουμε και όχι να παρεμποδίζουμε την έρευνα και την καινοτομία και την ανάπτυξη. Και χρειάζονται πολλές μελέτες για τα βιοκτώνα και τη συμπεριφορά του στο νερό. Γιατί μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ λίγα τα στοιχεία που έχουμε. Στόχος του παρόντος κανονισμού, λοιπόν, όπως σωστά λέγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς και πιο ταχεία διαδικασία και πιο ελαφρία, ε, όχι χρονοβόρα και βαριά. Αλλά Προς το παρόν αρμόδια για την αδειοδότηση είναι τα κράτη-μέλη. Και μόνο τα σχετικά κίνδυνα προϊόντα ε, θα ε, εμπίπτουν σε μια πανευρωπαϊκή έγκριση και αδειοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει θέλουμε να μειώσουμε το κόστος. Το υποστηρίζουμε αυτό, αλλά προς το παρόν δεν το βλέπω στην πρόταση της ενσωματωμένου. Είναι ε, τραγικά τα έξοδα αν θα πρέπει να ελέγχονται όλες οι δραστικές ουσίες. 3 με 5 εκατομμύρια ευρώ σημαίνει αυτό. Η ΕΧΑ ζητάει 400.000 ευρώ για να βάλει στο παράρτημα ένα, μια ουσία. Και για το προϊόν χρειάζεται τελικά 90.000 μέχρι 200.000 ευρώ. Σούμα τελικά 3,5 με 5,6 εκατομμύρια ευρώ για να βγάλεις μια ουσία και ένα προϊόν στο εμπόριο. Δεν ξέρω αν έχω κάνει λάθος στους υπολογισμούς και παρακαλώ την Επιτροπή να με διορθώσει ότι ερμηνεύω λάθος τα στοιχεία που κάνω ε, εδώ στην εκτίμησή μου. Αν ισχύει αυτό, αν είναι τόσο απαγορευτικό το κόστος όπως εγώ το υπολόγισα, ε, τότε ας μην εκπλησόμαστε που πολλές εταιρείε σταματούν την έρευνα και την ανάπτυξη. Τα βιοκτώνα είναι πολλά και έχουν και ειδικέ εφαρμογέ. Δεν είναι τόσο πολλά και τόσο μεγάλη η μάζα τους ε, και η χρήση τους όσο είναι τα φυτοφάρμακα, οπότε δεν είναι και κερδοφόρα τόσο πολύ. Οπότε σταματούν την έρευνα. Και τελικά θα χάσουμε ουσίες και έρευνα για λόγους ε, υψηλού κόστους και όχι όντως χαμηλού, χαμηλού κινδύνου. Τα κριτήρια που προτείνονται είναι σωστά, αλλά ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς είναι δυνατόν στο άρθρο 5 γάμα να μην ε, βάζει ε, εξαιρέσεις για τα φυτοφάρμακα. Ακόμα και αν ο κίνδυνος για το περιβάλλον ή την υγεία είναι μεγαλύτερος αν δεν συμπεριληφθεί μια δραστική ουσία. Ιδιαίτερα στην καταπολέμηση ε, κάποιων ζυζανίων ε, και, και νοσημάτων που μεταδίδονται με έντομα, ιδιαίτερα στην Νότια Ευρώπη, χρειάζεται ευρία παλέτα δραστικών ουσιών. Υπάρχει ο δάγκιος πυρετός, ε, ε, ο πυρετός τσιγκουνγκούγια που μεταδίδονται πούμε, με σκνήπες ή με κρότονες. Τι θα γίνει. Αυτό είναι πιο επικίνδυνο από ότι η χρήση των βιοκτώνων. Τα παράστα θα εμφανίσουν μεγαλύτερη αντίσταση και αντοχή στις ουσίες τελικά και αυτό θα έχει ολέθριες συνέπειες. 4 Φεβρουαρίου του 2009 πέρασε ένα ψήφισμα το Κοινοβούλιο για τη μελλοντική πολιτική του κλίματος και όλες οι πολιτικές ομάδες συμφώνησαν ότι υπάρχει ο κίνδυνος η κλιματική αλλαγή να ευνοήσει σημαντικά την εμφάνιση πολλών ασθενειών. Και στο άρθρο 159 γίνεται λόγος για τη σημασία ε, των ε, ε, ειδικών ενδυμάτων, χρησιμοποιούμε σπρέι, παρασιτοκτόνα, κουνουπιέρε κτλ. Με όλα αυτά θα εξαφανιστούν τα ε, τροπικά νοσήματα που βλέπουμε στην Νότια Ευρώπη ήδη να εμφανίζονται. Βλέπουμε την κλιματική αλλαγή και το έχουμε κατανοήσει ότι ε, κινδυνεύουμε και από ε, νοσήματα θερμών κρατών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει και για κάποια υλικά που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την προστασία του καταναλωτού και για την προστασία από του ανταγωνισμού. Στην Ευρώπη τα υλικά που κυκλοφορούν στο μέλλον θα πρέπει να ε, έχουν υποστεί επεξεργασία μόνο με τα βιοκτώνα που επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Μίλησε για μικητοκτόνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε παπούτσια και ε, επιπλά και που χρησιμοποιούνται στην Άπο Ανατολή και τι έλεγχος χρειάζεται. Τώρα, γίνεται μια πρόταση να υπάρχει σήμανση των ε, υλικών που έχουν υποστεί επεξεργασία με αναλυτική αναφορά άλλων των ουσιών. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι γεγονός ότι τα υλικά και τα προϊόντα στην παραγωγή τους θα πρέπει να έχουν ε, υποστεί επεξεργασία ε, με προϊόντα που επιτρέπονται και είναι αυστηρές οι διαδικασίες έγκρισης και θα πρέπει ο καταναλωτής να μπορεί να επαφείται. Και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα διαβατήριο ή με μια κάρτα βιοκτώνων και να γράφονται όλες οι ουσίες που έχουν χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή ή στην επεξεργασία του προϊόντος. Δεν νομίζω ότι βοηθάει αυτό. Τα βιοκτώνα χρήσιμα στην καθημερινή υγιεινή μας τα χρησιμοποιούμε όλοι. Είναι, επαναλαμβάνω, ε, ε, εκ των όνων στη ζωή μας. Με τη νέα πρόταση για τον κανονισμό έχουμε την ευκαιρία να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση και να περιορίσουμε τους κινδύνους. Ελπίζω Λοιπόν και προσβλέπω να έχουμε πολύ ε, καλή συνεργασία και προτάσεις από τους συναδέλφους και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κυρία Κλάς για την εκτενέστατη ευεριστατωμένη σας παρουσίαση και απάντηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τους κοιόδης τώρα εισηγητές από τις πολιτικές ομάδες. Ο Νταν Γιώργενσεν πρώτος. Thank Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επιτροπή και την κυρία Κλάς. Η κυρία Κλάς μίλησε εκτεταμένα και με πάθος για τις χαρές, τα θετικά των βιοκτώνων. Αναγνωρίζω ότι είναι σημαντικά τα βιοκτώνα και ότι έχουν πολύ χρήσιμες εφαρμογές ε, στην ε, σημερινή μας κοινωνία. Ωστόσο, η παρέμβασή σας περιείχε πολλά στοιχεία της ε, συζήτησης που είχαμε για τα παρασιτοκτόνα στην προηγούμενη θητεία μας. Παρατήρηση εκτός μικροφώνου η, η συγγήτρια λέει ναι, από εσάς εξαρτάται. Ε, ναι, πράγματι εξαρτάται και από μένα και από εμά. Ε, μπορώ να πω ότι ναι, τα βιοκτώνα είναι δώρο του κυρίου και δεν ε, χρειάζεται να κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Δεν θα το κάνω αυτό. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα βιοκτώνα είναι χημικά που χρησιμοποιούνται για να σκοτώσουν, να βλάψουν ή να αποτρέψουν ζωντανούς οργανισμούς. Αυτό θα πρέπει πάντα να το έχουμε κατά νου. Τα βιοκτώνα μπορεί να είναι και πολύ επικίνδυνα. Μπορεί να έχουμε πολύ σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον. Και γι' αυτό βρίσκω θετικό ότι η Επιτροπή δηλώνει ότι αυτός είναι ένας από τους μια από τις βασικές προτεραιότητες ε, της αναθεώρησης της ε, νομοθεσίας. Να πω ότι δεν θεωρώ ότι αυτό αντικατοπτρίζεται σαφώς στην πρόταση. Θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στο τι γίνεται για να μειώσουμε το κόστος και στο τι γίνεται για να βελτιωθεί το περιβάλλον και η προστασία της υγείας. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι η επικέντρωση του κειμένου είναι στο πρώτο και όχι στο δεύτερο. Μόνο τρει κουκίδε σε τρία σημεία υπάρχουν στην ε, προστασία του περιβάλλοντο, ενώ εννέα υπάρχουν ε, στις, ε, στη μείωση των δαπανών. Αν εξετάσετε και το περιεχόμενο των περιπτώσεων που αναφέρετε θα, πιστεύω ότι πολλοί θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι η ισορροπία δεν ευθυγραμμίζεται με την παρέμβασή σας. Ωστόσο, θα πρέπει να πω ότι υπάρχουν και πολλά θετικά στοιχεία στην πρόταση. Για παράδειγμα, βρίσκω εξαιρετικά θετικό ότι συμπεριλαμβάνονται τώρα τα επεξεργασμένα προϊόντα. Πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και ενδεχομένως θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συγκεκριμένη πτυχή ακόμα περισσότερο. Κάποιες από τις αδυναμίες που βλέπω έχουν να κάνουν με τη διατύπωση. Πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα να επικεντρωθούμε περισσότερο στην υγεία και στο περιβάλλον, όπως λέω εγώ. Η διατύπωση όμως στους ορισμούς, για παράδειγμα, είναι ιδιαίτερα αποδυναμωμένη. Όταν μιλάμε για, όταν έχουμε... όταν μιλάμε για τον ορισμό για τον χαμηλό κίνδυνο, η παρούσα διατύπωση, πιστεύω, ότι μπορεί να μην είναι επικοδομητική. Μακρηγορώ. Ναι, α, νόμιζα ότι, ε, ότι θεωρήσατε ότι ο κόσμος κάνει θόρυβο. Θα είμαι πολύ σύντομος. Πρόεδρος, έχουμε έξι παρεμβάσεις ακόμα και είναι έξι και τέταρτο. Θα έχουν μόνο δύο λεπτά ο καθένας. Ε, η κυρία Κλάς με προκάλεσε όμως. Ε, θέλω λοιπόν να αναφερθώ στον ορισμό για το χαμηλό κίνδυνο και τι κατευθυντήρες γραμμέ για την υποκατάσταση. Βρίσκω ιδιαίτερα ε, αδύναμα τα σημεία αυτά του κειμένου. ευχαριστώ Γιάννη. Κορίν Λεπά. δύο λεπτά. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ίσως καλό θα είναι να συνεχίσω στην ίδια γραμμή με τον προλαλήσαντα για να εφαρμόσουμε, να πω ότι τα βιοκτώνα είναι ένας άλλος ε, τρόπος να μιλάμε για ζανιοκτώνα, είναι όμως για ανθρώπινη χρήση και όχι για γεωργική χρήση και άρα θα έπρεπε να είναι αντικείμενο μιας ε, ακόμα πιο αυστηρής ε, νομοθεσίας, γιατί Για τα ζενιοκτώνα είναι πιο δικαιολογημένο γιατί μπορεί να πούμε ότι η γεωργία ίσως και να τα χρειάζεται, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Αν υπάρχουν σημεία τα οποία προοδεύουν σε αυτή την οδηγία, εγώ διαπιστώνω ότι όσον αφορά κυρίως τη διαφάνεια στην ενημέρωση υπάρχουν εξαιρετικά πολλές εξαιρέσεις που προβλέπονται και ότι θα πρέπει να έχουμε πλήρη και απόλυτη ενημέρωση του καταναλωτή για όλα τις αρνητικές δυνατότητες. Πιστεύω πως εδώ όλα αυτά είναι πολύ περιοριστικά σε σχέση με τον αριθμό εξαιρέσεων που προβλέπονται για αυτό το λόγο. Είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό αυτό και πιστεύω ότι θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο αυστηροί για τα είδη των προϊόντων και τον τρόπο έγκρισής τους, γιατί και πάλι οι συνέπειές τους για την ανθρώπινη υγεία υποτιμά, υποτιμάται υποτιμώνται μάλλον, σε σχέση με περιπτώσεις που έχουν ήδη προηγηθεί. Ευχαριστώ. Ήσασταν καταπληκτικοί και πολύ σύντομοι. Η Μισελ Ριβάζη. Πιστεύω ότι Βασικά για τα βιοκτώνα θα έπρεπε να είμαστε συνεπείς με την νομοθεσία για τα ζενιοκτώνα. Είναι το ελάχιστο γιατί είναι προϊόντα που είναι παρόμοια φύσης αλλά όπως είπατε ε, κυρία Κλάς αφορούν την ε, απολύμαση, την υγιεινή και θα πρέπει επίσης να, κάνουμε, να δούμε και τη σχέση κινδύνου με όφελος. Αν δεν υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις για τα προϊόντα τα οποία ε, περιέχουν τα βιοκτώνα για, κατά την άποψή μου υπάρχουν δύο πτυχές πολύ σημαντικέ και θα πρέπει να αναφερθούν κατά τη διάρκεια τη συζήτηση. Είναι η ευθύνη των κρατών μελών στην αδειοδότηση. Και το δεύτερο στοιχείο είναι τα κριτήρια συμπερίληψης για τις ενεργές ουσίες. Είναι δύο ε, στοιχεία για τα οποία έχουμε πολύ τσακωθεί για τα, ε, τη συζήτηση για τα ζενιοκτώνα και αν δούμε τις λεπτομέρειες για τα βιοκτώνα είμαστε πολύ πιο ελαστικοί και χαλαρή. Όσον αφορά την ευθύνη των κρατών μελών, υπάρχει δυνατότητα μη έγκριση για τα κράτη-μέλη, για τα ζυζανιοκτώνα. Δηλαδή, αν μια χώρα έλεγε Όχι, δεν σα δίνουμε την άδεια, το δεχόμασταν. Ενώ για τα βιοκτώνα θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά αμοιβή αναγνώριση. Αρκεί δηλαδή μια χώρα να πει Εμεί το αφήνουμε, το εγκρίνουμε, για να το εγκρίνουν και όλε οι υπόλοιπε χώρε. Για μα αυτό δεν είναι σωστό. Πάντοτε τσακωνόμασταν για την κυριαρχία των χωρών όσον αφορά την έγκριση τέτοιων βιοκτώνων ή ζυζανιοκτώνων. Πριν. Τώρα, οι όροι για τις ε, τοπικές περιστάσεις. Ένα κράτος μέλος ήταν ε, ε, ελεύθερο για να τροποποιήσει την νομοθεσία για τα ζανιοκτώνα, ενώ για τα βιοκτώνα χρειάζονται διάφοροι όροι να πληρούνται. Δυνατότητα χρήση. Για τα ζενιοκτώνα ήταν δυνατόν να περιοριστεί η χρήση σε σχέση με. αντίστοιχα για κάθε χώρα, ενώ για τα βιοκτώνα όχι. Δηλαδή, Βλέπετε, είναι απίστευτο για τα βιοκτώνα. Έχουμε πολύ λιγότερε δυνατότητε από αυτά που είχαμε καταφέρει σε σχέση με τα ζανιοκτώνα. Για την κεντρική αδειοδότηση. Για τα ζανιοκτώνα δεν ήταν δυνατόν. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα ζανιοκτώνο Κάθε κράτος έπρεπε να το εγκρίνει χώρια. Ενώ εδώ αυτομάτως γίνεται μια κεντρική αδειοδότηση για τα βιοκτώνα και για τα προϊόντα χαμηλού κινδύνου. Βρίσκω λοιπόν ότι για τα βιοκτώνα είναι πολύ πιο χαλαρή η κατάσταση, δηλαδή παραμελείται η ε, κυριαρχία των κρατών ενώ πρέπει να ενισχυθεί. Και θα πάω γρήγορα. Δεύτερον, τα κριτήρια αποκλεισμού για τις ενεργές ουσίες. Ορισμένα κριτήρια που ίσχυαν για τα ζεντοκτώνα δεν ε, προτείνονται για τα βιοκτώνα. Υπήρχαν ε, για τα επίμονα στοιχεία, τα βιοσιορευτικά, τα τοξικά. Όλα αυτά δεν υπάρχουν για τα βιοκτώνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ριβάζη, δεν έχετε άλλο το λόγο. να και τα λοιπά και αυτά θα πρέπει να σωματωθούν. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Φυσικά επιφυλάσσομαι να μελετήσω το κείμενο της πρότασης της Επιτροπής, αλλά βεβαίως και εκτιμώ την δυνατότητα κεντρικής έγκρισης φυσικά θα πρέπει να συνδέεται με τις εθνικές εγκρίσεις. Έπειτα θα πρέπει να υπάρχει και μια διαφορά ανάμεσα στην χρήση με απελευθέρωση υλικού και άνευ που θα μπορούσαν να ορίζονται διαφορετικά, να διέπονται από διαφορετικές νομοθεσίες. Υπογραμμίζω ωστόσο την ανάγκη να γίνεται μια έρευνα πολύ δραστηριά για τα βιοκτώνα γιατί οι συνθήκες αλλάζουν. Οι κλιματικές αλλαγές αντιστοιχούν και σε μια τροπικοποίηση του περιβάλλοντός μας. και θα πρέπει να έχουμε και βιοκτώνα που θα σταθούν στο ύψος των περιστώσεων. Υπάρχουν και έρευνες που αποδεικνύουν πως υπάρχουν βιοκτώνα τα οποία είναι πολύ επιλεκτικά και άρα μπορούν να έχουν ε, πολύ, πολύ περιορισμένες επιπτώσεις στο άνθρωπο. Και αυτό θα πρέπει να ευνοηθεί. Πάντως ευχαριστώ την κυρία Κλάς, ευχαριστώ την Κομισιόν και επιφυλάσσομαι να μελετήσω και πάλι. Μάλλον εις βάθος την πρόταση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριος Ρώση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να κάνω μια παρέμβαση για τι θέσει απασχόληση. Μπορώ να το κάνω σε σχέση με αυτό ή να σα δώσω. Μάλλον για την ημερήσια διάταξη, με συγχωρείτε. Ε, να το κάνω τώρα. Εγώ θα ήθελα να σας ζητήσω να αξιολογήσετε, να λάβετε υπόψη μάλλον, όταν υπάρχει τόση ύλη να εξετάσουμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε πολύ σημαντικά και λεπτά θέματα, θα πρέπει το Προεδρείο να ε, παρατείνει τις εργασίες για να μπορούν όλοι να παρεμβαίνουν αρκούντος γιατί δύο λεπτά για ένα έγγραφο 150-160 σελίδων που αφορά ένα τόσο λεπτό ζήτημα όπως η ανθρώπινη υγεία, νομίζω ότι υποτιμάται την, το θέμα. Λοιπόν, ή θα παρέμουν λιγότεροι ή θέλουμε περισσότερο χρόνο. Να πω τώρα για τις της Είναι ένα θέμα πάρα πολύ λεπτό, Πρόεδρε και συνάδελφοι, γιατί μπορεί να δημιουργήσουμε, αν είμαστε εξαιρετικά αυστηροί, να δημιουργήσουμε πολύ σοβαρά προβλήματα στους φορείς ε, στους, ε, του τομέα. Γιατί ε, εντάσσεται και η πρόταση που σχετίζεται με αυτές τις διατάξεις και λέει λοιπόν άρθρο τάδε της συνθήκης του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιοκτώνα. Ένα ένα αντικείμενο το οποίο εισάγεται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί ικανά εάν έχει υποστεί την ίδια κατεργασία όπως και τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Άρα λοιπόν καλό την Κομισιόν να εκτιμήσει σοβαρά ποια είναι τα μέσα που θα έχουμε στη διάθεσή μας στη συνέχεια για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τα όσα γίνονται εκτός Ένωσης. Γιατί αν εμείς επιβάλλουμε αυστηρούς κανόνες εντός Ένωσης και γι' αυτό συμφωνώ να επιβληθούν, ναι, αλλά να μην αλλά από την άλλη πλευρά δεν βρούμε επαρκές, επαρκές σύστημα ελέγχου, θα βλάψουμε τις δικές μας επιχειρήσεις χωρίς να εξυπηρετήσουμε όμως αντίστοιχα τους πολίτες μας. Ευχαριστώ, Ένια Βάισκερβερ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Κρίστα Κλάς για την ε, εισαγωγική της παρουσίαση ήταν εκτενέστατη και πολύ καλή. Στόχος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και αυτό είναι η απόλυτη έννοια μας και η φροντίδα μας ε, για την αναθεώρηση. Όπως είπε και ο δεν θα πρέπει ε, να δούμε τι γίνεται με την αδειοδότηση. Η παλιά όμως οδηγία για τα βιοκτώνα εμφάνισε πολλές αδυναμίες που δεν μπόρεσαν όλες να διορθωθούν και να βελτιωθούν. Υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία, μεγάλο κόστος για ελεγκτικές διαδικασίες, για αδειοδότηση και έγκριση. Μέχρι τώρα δεν είχαμε σχεδόν καθόλου, για να μην πω μηδενική τελείως έρευνα και καινοτομία και δεν έγιναν καθόλου βελτιώσεις. Δύο-τρία παραδείγματα. Πρώτον, στην πρόταση αυτή παραμένει γεγονός ότι τα βιοκτώνα ουσιαστικά ε, εγκρίνονται από τα κράτη-μέλη. Μόνο στα χαμηλού κινδύνου υπάρχει ευρωπαϊκή έγκριση. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι στόχος δεν θα πρέπει να είναι τελικά να έχουμε εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με ενιαία και μεγάλη προστασία. Και για το περιβάλλον βοηθάει αυτό και τα κριτήρια είναι τα ίδια, ενώ τώρα κάθε κράτος μέλος κάνει ό,τι του καπνίσει. Και επιπλέον, αν έχουμε και πολύ κακή αμοιβαία αναγνώριση που δεν λειτουργεί σωστά και δεν προβλέπεται με τρόπο επαρκή στην οδηγία, τότε δεν πρόκειται ποτέ να ενώσουμε την Ευρώπη σε αυτό το σύστημα. Αντίστοιχες συζητήσεις είχαμε στα φυτοφάρμακα, αλλά εκεί η πρόταση της Επιτροπής έλεγε τουλάχιστον ότι θα υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση, που ήταν ήδη πολύ μεγάλο βήμα προς την εναρμόνιση. Και τώρα ε, μου λείπει αυτό. Και ε, προς όφελος των ε, καταναλωτών, αλλά και των ε, προποθέσεων του ανταγωνισμού για τους μικρομεσαίους. Τώρα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, πολύ σύντομα, θα πρέπει να βρούμε μια λύση και ανάμεσα στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλες καταστάσεις όπως είναι τα πειραματόζα και για τα κριτήρια επιλογής ισχύουν τα ίδια και η ίδια συζήτηση με τα φυτοφάρμακα. Εγώ ενοχλούμαι πάρα πολύ όταν ξεφεύγουμε από το ρίσκο και μιλάμε για κίνδυνο. Στα καλλιντικά, ας πούμε, είχαμε άλλη προσέγγιση και θα προτιμούσα και εδώ το ίδιο να επιλέξουμε. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά για την Κομισιόν, αν θέλει. Κυρία Πούσκα συγγνώμη. κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θα είμαι πάλι πολύ σύντομη. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές ε, καθώς και τους άλλες βουλευτές που στηρίζουν γενικά την ε, πρόταση και τους ε, στόχους μας. Πράγματι η έμφαση δίδεται κυρίως στη μείωση του κόστους, αλλά αυτό δεν είναι εις βάρος του περιβάλλοντος, διότι τον περιβαλλοντικό στόχο τον πετυχαίνει ήδη η υπάρχουσα οδηγία. Αν λοιπόν ήταν πιο αποτελεσματική η υπάρχουσα οδηγία, θα είχε ήδη επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό ο στόχος μας ως προς την προστασία του περιβάλλοντος. Απλά κάνουμε δηλαδή πιο αποτελεσματικό το σύστημα και έτσι εξηγείτε πώς έχετε την εντύπωση και πώς βλέπετε περισσότερες κουκίδες, περισσότερες περιπτώσεις ε, όσον αφορά στο κόστος. Ε, αναρωτιέμαι ποιο έγγραφο είδατε, ελπίζω να μην ήταν οι σημειώσει μου. Ε, πάντως είναι σαφές Ε, αλλά ε, όπω είπαμε, αυτό δεν είναι, και όπω τόνισε και η κυρία Κλάσ, αυτό δεν γίνεται ει βάρο του περιβάλλοντο και τη προστασία ε, τη υγεία. Ο το, τομέα των βιοκτώνων ε, είναι ιδιαίτερα ποικιλόμορφο. Έχουμε ε, χημικά για τα πλοία, έχουμε απολυματικέ ουσίε, έχουμε ουσίε που χρησιμοποιούνται σε δημόσια πάρκα. Είναι, έχει τεράστια ποικιλομορφία ο τομέα αυτό. Και τα, τοπικά ε, χαρακτηριστικά είναι ε, λιγότερο σημαντικά από ότι στη γεωργία. Υπάρχουν δηλαδή ε, πρότυπα που μπορούν να εφαρμοστούν στο σύνολο της κοινότητας χωρίς να ληφθεί υπόψη ο τοπικός ε, παράγοντας. Δηλαδή, όπου είναι δυνατό θα πρέπει να επιδιώξουμε ευρωπαϊκή έγκριση και γι' αυτό επιλέξαμε ένα πιο ουδέτερο σύστημα έγκρισης. Θεωρήσαμε δηλαδή πιο κατάλληλο και προσαρμοσμένο στα διάφορα ε, χαρακτηριστικά του τομέα των βιοκτώνων. Μπορούμε βέβαια να το συζητήσουμε αυτό περαιτέρω. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την υποστήριξή σας ε, για τα ε, επεξεργασμένα προϊόντα και με το άρθρο για, τις, ε, για τα επεξεργασμένα υλικά. Ακριβώ αυτό θέλουμε να επιτύχουμε. Επίσης, ο ορισμός ε, για το χαμηλό κόστος είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε να προωθήσουμε την χρήση βιοκτώνων που είναι λιγότερα επικίνδυνα και θέλουμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίε επιχειρήσεις, διότι με την κεντρική διαδικασία είναι πιο εύκολο για τις μικρές επιχειρήσεις να ε, επιδιώξουν ε, την καινοτομία και την έρευνα για τέτοια προϊόντα, όπως τόνισε και ο κ. Πρόντι. Γενικά πιστεύουμε ότι τα βιοκτώνα είναι εξίσου σημαντικά ή ίσως ακόμα και περισσότερο σημαντικά από τα παραστοκτόνα με όλο το σεβασμό που τρέχω για τα παραστοκτόνα επειδή ακριβώς υπάρχει ε, η πτυχή της ε, δημόσιας υγείας για την, ε, όσον αφορά την απολύμανση κλπ. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι ο τομέας των βιοκτώνων είναι λιγότερο σημαντικός από τα παρασιτοκτόνα. Τα Χαρακτηριστικά όμως είναι διαφορετικά. Υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλομορφία στον τομέα αυτών ε, και περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάτσω μαζί με την κυρία Κλάς να κάνουμε λίγη αριθμητική μαζί. Δεν έχω κάνει τους υπολογισμούς όλους, αλλά είναι σαφές ότι το κόστος μπορεί να είναι υψηλό. Η πρόταση πάντως στοχεύει ακριβώς στη μείωση του κόστους και η περισσότερη παραγωγή είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτοί που διαθέτουν δηλαδή τα προϊόντα στην αγορά. Πολύ περισσότερο από ότι ε, στην περίπτωση των ε, επιχειρήσεων που παράγουν ε, τις ε, αρχικές ουσίες, τις δραστικές ουσίες, που συνήθως είναι μεγάλες χημικές επιχειρήσεις. Ε, αυτοί που δημιουργούν το τελικό προϊόν, λοιπόν, είναι συχνά μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η έγκριση των προϊόντων ε, στοιχίζει λιγότερο από ότι η έγκριση των δραστικών ουσιών. Νομίζω ότι έκανα τις βασικές παρατηρήσεις ε, για τις πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις που ακούσαμε και προσλέπω σε περισσότερες ενδιαφέρουσες ε, και επικοδομητικές συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Έξασα... Ξέχασα την κυρία Κέρλινγκ που είναι σκιώδης εισηγήτρια, αν έχετε ένα-ενάμιση λεπτό. εντάξει κύριε Πρόεδρε, δεν θα το πάρω προσωπικά. Έχω κάποιες παρατηρήσεις, ε, θα τις, θα τις ε, διαβάσω απευθείας στην κυρία Κλάς και έτσι θα τράξω την ευκαιρία να είμαι πρώτη στο κατάλογο των μιλητών στην επόμενη συζήτηση. Ε, είσαστε μεγαλόψυχοι. Κρίστα, έχεις κάτι να προσθέσεις? Διότι ήδη έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο μας. Ε, κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους, για τις παρεμβάσεις τους. Ε, το ήξερα βέβαια ήδη από πριν ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Προσβλέπω στην καλή συζήτηση. Νομίζω ότι σήμερα πολλοί καν δεν έχουν, δεν έχουν διαβάσει την πρόταση κανονισμού. Ε, προσβλέπω και στην ώρα της αριθμητικής με την Επίτροπη και ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε μια καλή κατεύθυνση, μια καλή προσέγγιση. πιστεύω ότι θα βρούμε μαζί μία λύση, διότι δεν διαφέρουν οι στόχοι μας. Μας ενδιαφέρει η υγεία, το, ε, τα στάνταρ υγιεινής κλπ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αν συμμετάσχει και ο Ντάν Γιούργενσεν θα είναι ακόμα πιο πλήρης, ε, θα είναι ακόμα πιο πλήρης το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ.